Donc, nous commençons notre réunion par l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons clarifier le point numéro 14. Madame Eva Joly est la rapporteure responsable, non pas pour un. Η κυρία Eva Joly έχει δύο νομοθετικά ψηφίσματα, όχι ένα. Ε, παρακαλώ, μην μιλάτε δυνατά. Συνεχίζουμε. Διαφωνείτε με το σχέδιο ημερήσια διάταξη όπω τροποποιήθηκε. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, les recommandations λοιπόν, συστάσεις και αποφάσεις των συντονιστών της 24 η Μαΐου θα εγκριθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση και περνούμε αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξη που αφορά την ανταλλαγή απόψεων ε, για την αναπτυξιακή πολιτική. Ξέρετε ότι η αναδιετή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταθέτει έκθεση ε, σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σε 12 συγκεκριμένους τομείς και η ιδέα είναι να συνεχίζουμε ε, τη βελτίωση βάσει των όσων συνιστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, η κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρσι το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση 2011 για τη συνοχή ε, των πολιτικών ή την ανάπτυξη και ως ήθιστε περιμένουμε ναι, εμείς να συνεισφέρουμε υπομορφή ε, έκθεση πρωτοβουλίας από την εισηγήτριά μας που είναι η κυρία Μπίργκιτ Σνίμπερ Γιάστραμ, διαρκής και μόνιμη εισηγήτρια και θα μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία της έκθεσης. Δίνω αμέσως στο λόγο στην κυρία Σνίμπερ Γιάστραμ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε και πάλι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην αναπτυξιακή συνεργασία, όπως είπατε και εσείς, και αυτή είναι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Κατά την περασμένη διετία είχα μέτρητες συζητήσεις και είχα την ευκαιρία να συλλέξω πολλές εμπειρίες για την τελική έκθεση, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ε, επί της αρχής, καταρχάς, η ονομασία είναι κάπως περίπλοκη και ιδιαίτερα τεχνική ίσως. Φοβάμαι ότι δεν αλλάζει δυστυχώς τώρα τίποτα σε αυτό, αλλά θα πρέπει πάντα να ξεκαθαρίζουμε περί τίνος πρόκειται σε αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι πώς ε, θα κάνουμε την πολιτική μας βιώσιμη και αηφόρο. Αυτή είναι μια πολιτική του μέλλοντος, λοιπόν, η συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Και εδώ υπάρχει ένας ειδικά τεχνικός λόγος η αναπτυξιακή συνεργασία που κανονικά σε λίγο θα καταστεί τί, η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να είναι φόρ. Δηλαδή, όταν έχουμε πολιτικές ε, συνεργασία με άλλες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα πιο φτωχές θα ε, πρέπει να ε, διατηρηθεί η συνοχή της πολιτικής. Μόνο με μια τέτοια συνεκτική πολιτική μπορεί να έχουμε εταιρική σχέση ε, με τις χώρες και επί όρες. Και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε και τις πρώτες ύλες και τις νέες αγορές της Αφρικής και όχι αντίστροφα. Μόνο έτσι λοιπόν με την ε, συνοχή μπορούμε να ε, συνεχίσουμε με θετικέ πολιτικές και να ξεφύγουμε από αρνητικέ πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας. Μόνο με την αναπτυξιακή πολιτική λοιπόν και τη συνοχή της θα δημιουργήσουμε τι προποθέσει έτσι ώστε οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες των χωρών ΑΚΕ να έχουν την ευκαιρία και την ευθύνη να ε, επιτυχάνουν μόνοι τους επιτέγματα. Έχει αναγνωρίσει η Δανική Προεδρία αυτή τη σημασία και αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν το έχουν καταλάβει όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το προηγούμενο Σαββατοκυριακό είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στη Δανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά, ήδη και θα πρέπει να το πούμε και στην έκθεση. Αλλά Υπάρχουν κάποια θέματα πάρα πολύ περίπλοκα και δεν εντάσσονται σε όλες τις πολιτικές, δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο και πάντα θα πρέπει να ε, εκφράζουμε την κριτική μας για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, πολιτική συνοχή. Ε, γιατί αυτή είναι η θεσμοθέτηση της κριτικής, δηλαδή η αναγωγή της κριτικής σε θεσμικό επίπεδο. Έχετε ένα έγγραφο εργασία σήμερα στα χέρια σας Είχε ζητήσει κάποια άλλη επιτροπή να αναβληθεί ε, για λόγους ε, χώρου και έκθεση της έκθεσης δεν κατάφερε να επεκταθώ. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο σε ένα τόσο ευρύ πεδίο να συμφωνήσουμε. Κάποιος θα ήθελε ας πούμε να γίνεται εκτενέστερη αφορά σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ή άλλοι ε, θέλουν να βγουν ε, να εξαιρεθούν οι ε, κρατικές προμήθειες. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας νομίζω και για τα βασικά θέματα έχουμε συμφωνία. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η ισορροπία ανάμεσα σε θέματα ουσίας ε, περιεχομένου δηλαδή και της θεσμικής λειτουργίας. Τα θεσμικά ζητήματα ε, στην Επιτροπή ε, θα τα συζητήσω εκτός εκθέσεως ειδική συνεδρίαση με τους συντονιστές. Πάντως έχει καταστεί σαφές το εξή στην προηγούμενη διετία, ότι το βασικό πρόβλημα είναι πώς θα γεννηθεί, πώς θα προκαλέσουμε και θα δημιουργήσουμε την πολιτική βούληση για μια τέτοια πολιτική. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύνολο της εξωτερικής μας πολιτικής, γιατί μόνο έτσι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής θα είναι δεδομένη σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Αλλά το θέμα είναι τόσο περίπλοκο και χρειάζεται και τόσο πολλή συζήτηση και εκείνους που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική που υπερβαίνει κατά πολύ την έκθεση που τα αναφέρει ε, επιγραμματικά. θα πρέπει να πούμε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μας ακολουθούν σε αυτή την προσπάθεια ε, τις τροπολογίες θα σας τις στείλω ταυτόχρονα με το σχέδιο έκθεσης για να ε, αποφύγουμε επικαλύψεις και διπλές ε, αναφορές. Περιμένω με χαρά τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, εξ ε, του δικού μας σκιώδου ε, του κυρίου Πατρίστη Ρολιά λόγω των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία που σιάζει. Θα ήθελα καταρχά να εκφράσω την ικανοποίησή μας στην συγγήτρια για το βασικό άξονα που δίνει στην πολιτική ανάπτυξη. Το άρθρο όμω 208 της Συνθήκης Λισαβόνα είναι αρκετά φιλόδοξο και θα εξακολουθούν να είναι τεράστιες οι προσπάθειες που χρειάζονται. Γι' αυτό ελπίζουμε στην τέταρτη διετή έκθεση το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για το κόστος ε, που έχει η έλλειψη της συνοχής στις πολιτικές μας. Το έγγραφο είναι ε, εξαιρετικό, εκφράζει τις προκλήσεις η και για το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για τις επιμέρους πολιτικές. Η ομάδα μας έχει να κάνει κάποια σχόλια. Πρώτον, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας γιατί μέχρι σήμερα μόνο δύο άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν γνωμοδοτήσει για τη διετή έκθεση. Κρίμα που η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν έχουν ε, γνωμοδοτήσει, γιατί είναι μεγάλη σημασία του στην ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, συμφωνούμε με την πρότασή σας να δημιουργηθούν ε, ε, συγκεκριμένα σημεία στις αντιπροσωπείες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να ε, πάμε πιο πέρα. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ας πούμε, στα στρατηγικά σχέδια και ε, περιλαμβάνονται και κεφάλαια για άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει αυτή ανάλυση και για να συμφωνούμε με το άρθρο 12 της Συνθήκης του Κοτονού θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση και στρατηγικά έγγραφα για τις πολιτικές μετά από ευρύτατη συζήτηση και δημοκρατική με τις κοινωνίες, τα κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών στις εκάστοτε χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να αξιολογεί την κατάσταση και να δίνει με παραδείγματα τις επιπτώσεις της αναπτυξιακής πολιτικής σε λόγο χώρες. Καλωσορίζουμε μεν την ατζέντα για την αλλαγή η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ναι, μήπως θα μπορούσατε να τα λέτε με λιγότερο ηλικιώδη ταχύτητα. Μάλιστα. Θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι Μπορεί να καλωσορίζουμε, λέγω, την ατζέντα για την αλλαγή, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι ποτέ υποκατάστατο άλλων ε, υφισταμένων ρυθμιστικών πλαισίων και κανονιστικών πλαισίων σε μελλοντικέ αναπτυξιακέ πολιτικέ. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστή η Συμφωνία τη Κοτονού. Σε ό,τι αφορά τι επιμέρου κλαδικέ πολιτικέ που μπορεί να έχουν μεγάλη επίπτωση στην ανάπτυξη, θα θέλαμε να προσθέσουμε το εξή. Πρώτον, η ομάδα μα θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει η εφαρμογή της αρχής τη διαφοροποίησης να μην είναι αμυγής οικονομική λογική. Παράδειγμα, κανόνες για την εφαρμογή ε, μέσου χρηματοδότησης ε, και τη ανάπτυξη. 11 χώρες ε, της Λατινικής Αμερικής βγαίνουν από τη διμερή ε, συζήτηση, ενώ κάποιες ε, άλλες θα δουν τη βοήθεια να μειώνεται ή να καταργείται τελείως. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όχι μόνο το κατακεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και ο δείκτης ευαλωτότητας της οικονομίας και της ανάπτυξης, γιατί υπάρχουν χώρες που εξαρτώνται από την κλιματική αλλαγή και από λίγα προϊόντα στην παραγωγή τους. Η ε, εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την αναπτυξιακή πολιτική. Η μεταρρύθμιση των συστημάτων, ε, συστημάτων γενικευμένων προτιμήσεων ε, μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλές καταστάσεις. Χώρες με μέσο εισόδημα ή υψηλό μπορεί να χάσουν ε, την ιδιότητα της χώρας που εντάσσεται στη συνεργασία και είναι αυτό ένα στοιχείο που μπορεί να έχει επιπτώσει σε εξαγωγές του. Ανεργειακή πολιτική. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες ύλε για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αλλά αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις και το ξέρουμε. Η ε, ανεξέλεγκτη ε, εκμετάλλευση και η άναρχη όχι μόνο θα εξαντλήσει τις ε, πηγές αλλά θα ε, μειώσει και ε, τις ευεργετικές επιπτώσεις που έχουν σήμερα τα τροπικά οικοσυστήματα στους ντόπιου ε, πληθυσμούς. Και όχι μόνο στον πληθυσμό, αλλά και στις επιστησικές καλλιέργειες. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και επίγον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει αξιόπιστα στοιχεία για την αλλαγή της χρήσης γης και συγκεκριμένα οι καλλιεργήσιμες γης να χρησιμοποιούνται για παραγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης η μετανάστευση των ε, εργαζομένων θα πρέπει να μας απασχολήσει για να μην ε, πληγούν από διαρροή εγκεφάλων οι χώρες αυτές. Ελπίζουμε και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με την συγκήτρια προς την κατεύθυνση αυτή και σας ευχαριστώ. Οπότε, προτού δώσω τον λόγο στον συνάδελφο, θέλω να τον καλωσορίσω, διότι αντικατέστησε την κυρία Κέλλερ που πήγε στην Ίντα. Είναι ο κύριος Κιθ Τέιλορ, στον οποίο δίνω αμέσω τον λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, αντικατέστησα την ε, κυρία Κέλλερ, τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το πράξω στο μέτρο του δυνατού. Και ε, η ΣΚΑ και εγώ ουσιαστικά ανταλλάξαμε θέσεις. Ε, έλαβε τη θέση μου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και εγώ τη δικιά της εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, έπεσα κατευθείαν σε αυτό το πολύ βασικό θέμα και πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία διότι δεν είναι μόνο το ίδιο τραγούδι αλλά και τα ίδια λόγια του τραγουδιού δηλαδή πρέπει να εντοπίσουμε τις δυνατότητες του τι είναι δυνατόν να προσθεθεί στο κείμενο αυτό πράγμα που μόνο ένα έγγραφο εργασίας μπορεί να πράξει πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και εάν οι συστάσεις δεν ληφθούν υπόψη ή ε, αν δεν υπάρχει συνεκτικότης για ανάπτυξη και αυτή εμποδίζεται από τις ε, ε, διαφορετικές και αντιφατικές πολιτικές δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεπή πολιτική ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να δούμε σαν κοινοβούλιο πώς εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δικιά μας συνεκτικότητα για την ανάπτυξη και ε, αναφέρομαι εδώ παραδείγματο χάρη εις το διεθνές εμπόριο όπου ορισμένες αποφάσεις ε, ε, και τα θέματα για το GSP, για το ε, ε, για διάφορα θέματα ε, ή για το γεγονός ότι ευάλωτες οικονομίες δεν πρόκειται να βοηθηθούν από την Ευρώπη και αποκλείονται με, μου δημιουργούν προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να εκμεύσουμε τη σωστή πολιτική βούληση εάν θέλουμε η ίντα να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις και την ε, συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Γι' αυτό και θέλω να αναφερθώ εις ε, τις προτάσεις της ε, κυρίας Κέλλερ, δηλαδή να βελτιώσουμε τον μηχανισμό ο οποίος θα αποτελέσει το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα μας αποφύγει την προσπάθεια ε, διατυπώσεως εκθέσεων που αναφέρονται στην έλλειψη συνοχής αντί για τη συνοχή όπως ε, σήμερα και Γι' αυτό νομίζω ότι όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω το πρόγραμμα αυτό να μπορέσει να προωθηθεί ως το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Λεύιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Κιθ που αντικατέστασε στη ΣΚΑΛ. Θέλω και εγώ να προσθέσω λίγα σχόλια. Στο έγγραφο εργασία τη εισηγήτριά μα. Το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Αλία, ε, η οποία συντάσσει μια γνωμοδότηση. Και με μεγάλη ικανοποίηση παρατήρησα ότι η εισηγήτρια αναφέρει τις τρεις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν την ε, μεγαλύτερη επίπτωση ε, στι αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι το εμπόριο, η γεωργική πολιτική και η αλληλευτική πολιτική. Και αν διαβάσετε την έκθεση της ε, Κομισιόν, θα δείτε ότι πολλές σελίδε αναφέρονται στη μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής πολιτικής που θα μας εξασφαλίσει και επιστημιστική ασφάλεια. Ξέρετε ότι με την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής υπήρξαν κάποια προβλήματα τα τελευταία 6-7 χρόνια και μία από τις συνιστώσεις που θα πρέπει να απλουστευτεί πολύ περισσότερο ε, σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική είναι η λεγόμενη τομεακή στήριξη. Γιατί υπήρχε έλλειμμα στη δυνατότητα απορρόφησης των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει δηλαδή πόσοι αλία θέλουν να έχουν οι χώρες και δίνει κάποια χρήματα που συνοδεύουν ουσιαστικά τις αλληλευτικές συμφωνίες για να εξασφαλίσει την τομεακή στήριξη. Βασικά είναι βοήθεια. Και με αυτή τη βοήθεια ε, προσπαθούν στις τρίτες χώρες να δημιουργήσουν εθνικές αλληλευτικές πολιτικές. Αλλά ξέρουμε τώρα ότι πολλά από αυτά τα κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως θα έπρεπε Ξέρουμε ότι το δυναμικό απορρόφησης δεν ήταν επαρκές. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική να συντονίζεται με την αληθική πολιτική ως προς αυτό. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η αναπτυξιακή μας πολιτική. Δεν μπορεί να έχει συνεκτικότητα, συνοχή. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Τέιλορ, το μόνο που θέλω να προσθέσω για να συμπληρώσω είναι ακριβώς αυτό που ακούσατε από μένα μόλις τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε η μοναδική, το μοναδικό όργανο σε διεθνές επίπεδο που μιλάει για την συνοχή των πολιτικών μας. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, σε σχετικούς, με σχετικούς όρους, γιατί αν δούμε τι γίνεται και αλλού, είμαστε οι μόνοι που προβληματιζόμαστε σε αυτό το θέμα. Έπειτα, τα πάντα ρί, ο κόσμος αλλάζει και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Το θέμα είναι να δούμε αν προσαρμοζόμαστε με τρόπο συνεπή, με βάση τις δικές μας αρχές, ε, σεβόμε τις δικές μας αρχές, με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε, με κάθε ειλικρινία. Τρίτον, η βάση των δράσεών μας είναι η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Αν θέλουμε να σπρώξουμε περισσότερο την, και να προωθήσουμε τη συνοχή των πολιτικών, θα πρέπει όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι θεσμικοί φορείς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνταχθούν γύρω, πίσω από τις αρχές όπως προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Συνένεση. πρώτα στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια μπορούμε να καλέσουμε την ε, Λέδη Άστον για να προσυπογράψει και αυτή το ευρωπαϊκό έγγραφο ε, για τη συνένεση, την ευρωπαϊκή συνένεση. Νομίζω θα ήταν ένα καλό μήνυμα μέσα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά, αποτελούμε αραγές μέτωπο όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς. Ότι αυτή την αρχή όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς δέχονται αυτή την συνένεση του 2005. Στο μεταξύ βέβαια ε, έχει τροποποιηθεί η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ε, τροποποιήσουμε και ας προσαρμόσουμε αυτή τη συνένεση ε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κάτι που δεν υπήρχε το 2005. Έπειτα, τρίτη παρατήρηση, μέθοδος εργασίας μας. Πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί νομίζω κάθε χρόνο θα πρέπει να βλέπουμε όλες τις πολιτικές. Εντάξει, καλό είναι, αλλά σε κάποια θέματα καλό θα ήταν να σταθούμε περισσότερο. Παραδείγματο χάρη, να αναλύσουμε την επίπτωση της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Να έχουμε νούμερα, ποσοτικά στοιχεία. Να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Ποια ήταν τα θετικά και ποια ήταν τα αρνητικά. Από το 2000 μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν πολλά υπάρχει καλύτερο συντονισμό της αναπτυξιακή πολιτικής, αλλά και της κοινή γεωργικής πολιτική. Ιδίω για τα ποσά που αφορούν τις εξαγωγικές επιστροφές, που διαιρέθηκαν δια 30, αν δεν απατώμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αυτά τα ποσά. Πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν μπορεί να κάνουμε συνέχεια τα ίδια λογίδρια. Δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο γενικόλογοι πάντα. Ας έχουμε και τα μέτρα ε, για να προσμετρήσουμε την πρόοδο ή την αποτυχία. Το ίδιο και για το εμπόριο. Αν δούμε το εμπόριο ένα θέμα, θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση των ασθενών των τρίτων χωρών στα, στα γενώσιμα φάρμακα, στους, στα φάρμακα για το AIDS, τους αντιρετροϊούς. Ας μην είμαστε γενικόλογοι μόνο. Μονίμως α, αμφισβητούμε τα όσα έχουμε κάνει. Μήπως να δούμε και τα θετικά και μάλιστα με νούμερα, ποσοτικά, ούτως ώστε να προτάξουμε το συνεπή μη χαρακτήρα των πολιτικών μας και να συγκρίνουμε τις δικές μας πολιτικές με των υπολείπων, των άλλων, που δραστηριοποιούνται και αυτοί στην αναπτυξιακή πολιτική. Ούτως ώστε να δούμε σε σχετικούς όρους τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε χειρότεροι, το πιστεύω, ειλικρινά το λέω, δεν το πιστεύω νομίζω ότι θα πρέπει να συγκριθούμε με άλλους. Γίνεται αυτό. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις. Μελέτες, κοντραμελέτες, ε, μελέτες επιπτώσεων. Ε, στο έγγραφό μας, Agenda for Change, ε, πρόγραμμα δράσης για αλλαγή, Νομίζω ότι θα πρέπει με, βάση τα νούμερα, με βάση κάποια ποσοτικά στοιχεία, να απεικονίσουμε την πραγματικότητα. Για να δούμε αν υπάρχει συνοχή. Για να δούμε αν είμαστε πολύ, έχουμε μία έτσι, προσέγγιση πολύ χρηστική. Προσπαθούμε συνέχεια να εξηγήσουμε τι κάναμε στον τομέα της ανάπτυξης σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που έφερε για μας. Εντάξει, στο εμπόριο χρειάζονται και αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι συχνά ε, η βοήθειά μας δίνεται αμερόληπτα. Δεν είμαστε πάντα ιστερόβουλοι. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η Κομισιόν. Η κυρία Λομπιέσοβα. Euh, euh, Ευχαριστώ. Να απαντήσω στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Άκουσα την παρουσίαση με μεγάλο ενδιαφέρον. Χαίρομαι που πολλά από τα συμπία που εμείς προσπαθούμε να προτάξουμε στην έκθεση του 2011 ε, τα προτείνει και το Κοινοβούλιο στα πιο σημαντικά. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κρίμα που δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε ποσοτικά το πώς πήγαν οι προτεραιότητές μας τα τελευταία χρόνια. Μερικέ φορέ ε, δεν είχαμε τα αριθμητικά στοιχεία τη στιγμή που γράφαμε την ε, έκθεση. Προσπαθούμε να έχουμε περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και ελπίζουμε να κάνουμε περισσότερες συγκρίσει ε, στην έκθεση του 2013. Όλη η προσπάθεια μέτρησης, εφόσον δεν έχουμε κοινή μεθοδολογία, καθίσταται δύσκολη γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε τι έγινε και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν έχουμε όλη την ίδια μεθοδολογία, δεν θα είναι συγκρίσιμα τα νούμερα. Αυτή είναι μια πρόκληση και θα πρέπει να την εντοπίσουμε. Για τα υπόλοιπα σημεία τώρα. Έχω την εντολή να σας ξαναπώ ότι οι αρχές της συνοχής για την απτυξιακή πολιτική ε, υπάρχουν και στη συνένεση. Η συνένεση δεν έχει ξεπεραστεί από το πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, από το Agenda for Change. Και οποιοδήποτε σχέση το αντίθετο τον διαψεύδω. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε περισσότερο με τη συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική στην ατζέντα μας. Ε, γιατί δεν θέλουμε να ξαναμφισβητήσουμε τις ίδιες αρχές που υπάρχουν ήδη στη συνένεση. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ για τις αντιδράσεις σας. Ευχαριστώ. Euh, Η επόμενη ομιλήτρια δεν είναι εδώ. Η συγγήτρια για τα καταληκτικά της σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, σχετικά με την ε, πρόταση και τις κριτικές τη σημειώνω διότι εδώ πρόκειται για ένα έγγραφο εργασίας δηλαδή υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία ακόμη πρέπει να γίνουν αποδεκτά και εδώ ε, αναφέρουμε στο θέμα των focal points των αντιπροσωπιών Προσπάθησα να είμαι σύντομη λόγω του χρόνου, αλλά η αντιπροσωπεία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ε, για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά χρειάζεται και ε, ε, χρειάζονται και περισσότεροι πόροι και περισσότερο δυναμικό. Βεβαίως τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα ιδίω στα πλαίσια της πωλήσεως των όπλων πρέπει να τονιστούν και το Συμβούλιο αναφέρεται στο Country Level Dialogue το οποίο είναι κάτι ευπρόσδεκτο αλλά εδώ θα πρέπει να βρούμε μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση και τέλος θα τελειώσω με το τελευταίο σημείο λέγοντας ότι χρειαζόμαστε ε, μία πλήρη επάνδρωση της ε, BCD ε, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος. Δηλαδή η συζήτηση δεν πρέπει μόνο να γίνει τώρα αλλά και στο μέλλον και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα. Ευχαριστώ κυρία Χέστραμ και τώρα θα υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως αφενός Κολομβίας και Περού από την άλλη. Ο κύριος Πίνο Αρλάτσι, εάν έτσι προφέρετε το όνομά του, λυπάται που δεν θα παραστεί και ο κύριος Ρικάρντο Κορτές Λάστρα θα παρουσιάσει ανταυτού την πρόταση γνωμοδότησης και του δίνω τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Αρλάκη, ο εισηγητής ε, συντάκτη της καλύτερα απουσιάζει και ζητάει συγγνώμη. Ο κύριος Σαλάκη θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας και Περού είναι εκ των όνων για να ε, βελτιωθούν όσο γίνεται οι σχέσεις με τις χώρες αυτές. Ωστόσο, στη γνωμοδότηση ε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που μας ανησυχούν κάπως. Ιδιαίτερα αυτό που έχει να κάνει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να τονίσουμε τα εξή δύο σημεία. Πρώτον, η συμφωνία αυτή προϋποθέτει μια, ένα σαφές πλαίσιο και προβλέψιμο για να υπερβούμε αυτές τις ανησυχίες και με τις δύο χώρες αυτές. Έχουμε μπει σε μια δυναμική απαιτήσεων Τέτοιε απαιτήσει δεν έχουμε όμω από την Κίνα, το Ουσμπεκιστάν, τη Γουατεμάλα ή το Ελσαλβαδόρ, όπου συνάψαμε αντίστοιχε συμφωνίε και το Κοινοβούλιο ανέκαθεν εξέφραζε την ανησυχία του και για τι χώρε αυτέ ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό. Δεύτερον, η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην Κολομβία και στο Περού να ε, παίζουν με ίδιους όρους ε, διεθνώ με άλλε χώρε που έχουν τι ίδιε διευκολύνσει. Τουρκία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Ισραήλ. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η Κολομβία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες εκεί. Έχει ε, εγκριθεί ε, ε, ο νόμος για την αποκατάσταση των θυμάτων και την επιστροφή των γεών. Έχει κλείσει το διαβόητο ΝΤΑΣ. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει ενεργά στην εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων που θα υποχρεώνουν όλα τα μέρη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους. Θα ήταν καλό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κάποιους μηχανισμούς έτσι ώστε οι οικονομικές συμφωνίες και εμπορικές συμφωνίες να σημαίνουν ε, πραγματικές προόδους, ανθρώπινα δικαιώματα, σε δικαιώματα των εργαζομένων και άλλα. Αλλά όχι επιπλέον επιβαρύσεις και απαιτήσει ε, για μονομερή ε, αναστολή της συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά πηγαίνουν σωστή κατεύθυνση. Θεωρεί επίσης ο εισηγητής ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξακολουθεί να παρατηρεί στενά ε, την ε, υλοποίηση και την εκτέλεση των συμφωνιών και θα πρέπει με τρόπο διαφανή όσο και αποτελεσματικό να εφαρμόζεται η συμφωνία. Ζητεί λοιπόν από την αρμόδια επιτροπή ο εισηγητής να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία σε περίπτωση ε, της Λατινικής Αμερικής αυτό επιτρέπει να ε, αυξηθεί η στρατηγική μας συνεργασία με την περιοχή που είναι από τις περιφέρειες του κόσμου εκείνες που μοιάζουν περισσότερο με την Ευρώπη και πολιτιστικά και πολιτικά. Αυτό το είδαμε και με την έγκριση την περασμένη εβδομάδα ε, των 27 της Συμφωνίας αυτής ελεύθερων συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μέσνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κορτές που αντικαθιστά τον εισηγητή των συνδικαλιστών. όντως υπάρχει μια μακριά προϊστορία ε, στην έκθεση αυτή ε, και στην αρχή ε, υπήρχε μια ενεργή, συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία η οποία όμως μετά είχε τονίσει και τώρα υπάρχουν συμφωνίες μόνο με την Κολομβία και το Περού και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και γνωρίζω ότι εδώ ορισμένε ε, ε, πολιτικές ομάδες ε, έχουν αμφιβολίες αν όλα θα εξελιχθούν καλά με τις συμφωνίες αυτές και η αλλαγή όμως κατά άλλους επιτυγχάνεται μέσω του εμπορίου και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ε, λάβει υπόψη της αυτά τα θέματα και συγχρόνως να σκεφτούμε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και υπάρχει και μία ρήτρα η οποία επιτρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία αυτή σε άλλες χώρες, πράγμα το οποίο είναι προσόν για την περιοχή και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιληφθούν σε ψηφίσματα για να ενθαρρυνθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι ενδεχόμενοι υποψήφοι. Και εγώ είμαι υπέρ του να στηριχθεί εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος. Ευχαριστώ και δίνω τώρα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον κύριο Μικαλάντζελο Μαργκέρτια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια τα οποία απευθύνατε σχετικά με αυτή τη συμφωνία διότι όντως έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες επ' αυτού και με τα μεγάλης χαράς πρέπει να σας δώσω μία πρώτη ένδειξη για την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διάφορα έγγραφα τα οποία κυκλοφορούν στις Επιτροπές και κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει μία εξαιρετική διάσταση στην συμφωνία αυτή σχετικά με το πώς αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει ε, την ε, Κολομβία και το Περού να αναπτύξουν την ε, οικονομική τους πολιτική. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το διαπραγματευτήκαμε πάρα πολύ σκληρά κατά τα δύο χρόνια των διαπραγματεύσεων και είμαι βέβαιος ότι η συμφωνία αυτή είναι καλή. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό διότι ξέρουμε ότι η συζήτηση αυτή υπήρξε πολύ ε, έντονη και στο Κοινοβούλιο αλλά και έξω από εδώ, δηλαδή στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι διατάξεις που περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή σχετικά με ε, την διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών, τα περιβαλλοντολογικά δικαιώματα, τη δυνατότητα καταρτιστεί ένα σύστημα διαιτησίας και να περιλαμβάνει και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συμφωνηθεί και εδρεωθεί. Όσον αφορά τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο μία ρήτρα που υπάρχει σε άλλες συμφωνίες, αλλά για πρώτη φορά σε εμπορική συμφωνία πλαίσιο για πρώτη φορά ενώ υπάρχει στις συμφωνίες πλαίσιο εδώ σε μία εμπορική συμφωνία προβλέπεται ότι μπορούμε να άρουμε και να διακόψουμε είτε το σύνολο ή όλες τις, τις δυνατότητες συνεργασίας εάν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ ε, έντονα, ιδίως όσον αφορά ε, την, ε, τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών που είναι μη, κάτι το υποχρεωτικό. Οι χώρες αυτές πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών αν δεν έχει ήδη εδρεωθεί ο θεσμός και καλούμε όλους τους συμμετέχοντες και τους εμπλεκομένους στην κοινωνία των πολιτών να εκφραστούν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντολογικά δικαιώματα και ε, να μεταδώσουν τις απόψεις αυτές στους Ευρωπαίους ομολόγους τους που θα ε, είναι ένα πολύ βασικό θέμα όσον αφορά την ε, αναφορά της συμφωνίας. Υπάρχουν και άλλες μελέτες ε, και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ε, πρόσβαση και εξοικονόμηση δασμών μεταξύ μισού και ενός δισεκατομμυρίου ε, ευρώ ετησίως που θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κολομβίας και Περού και 1% του ΑΕΠ ή σχεδόν 1% του ΑΕΠ ε, θα, ε, θα αυξηθεί στις χώρες αυτές, ε, κάτι λιγότερο για την Κολομβία, κάτι περισσότερο για το Περού. Και αυτά είχαμε να ενημερώσουμε και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κορτές για να καταλήξει και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι για αύριο 5 Ιουνίου στις 12 ακριβώς. δεν θέλει το λόγο ο μιλητής, οπότε τώρα περνάμε στην ε, παρουσίαση του κυρίου Τάις Μπέρμαν που θα παρουσιαστεί από τον κύριο Λόζε, διότι ο κύριος Μπέρμαν δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Όπως ξέρετε είναι εισηγητής της Επιτροπής μας για την νομοθετική ε, έκθεση σχετικά με ε, την αναπτυξιακή πολιτική μέχρι 2014-2020 που προβλέπει χρηματοδότηση στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης. Το πακέτο αυτό καταρχήν θα εξεταστεί από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κοινό κανονισμό για όλες τις εξωτερικές δράσεις, πράγμα το οποίο έχει νόημα διότι οι περισσότερες λειτουργίες είναι ταυτόσιμες και συγχρόνως αυτό δίνει εξουσία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και ο εισηγητής είναι ο πρόεδρός της κύριος Έλμαρ Μπρόκ. όλα αυτά όμως είμαστε συνδεδιασμένη επιτροπή για όλες τις πτυχές που αναφέρονται αποκλειστικά ή ιδίως στην αναπτυξιακή συνεργασία και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Λόιζερ ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπέρμαν, ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον κύριο Μπέρμαν που είναι εισηγητής για την αναπτυξιακή συνεργασία και το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία το DCI. Υπάρχει στενή σχέση με το CIR. Γι' αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να, να ορίσει τον κύριο Μπέρμαν για την σύνταξη μιας γνωμοδότησης ε, που συμφωνήθηκε μαζί με την ΑΦΕΤ, γιατί είναι οι συνδυασμένες επιτροπές, δηλαδή είναι οι επιτροπές που εμπλέκονται και αυτές με βάση το άρθρο 50 θα πρέπει όλο το προσωπικό των επιτροπών να βοηθήσει τους εισηγητές για τους κανονισμούς ε, που αφορούν το CIR, αλλά και τις διατάξεις ε, του CIR που θα επηρεάσουν τα διάφορα μέσα. Αυτές οι συνεδριάσεις έχουν λάβει χώρα και ήταν πολύ θετικές, πολύ επικοδομητικές. Το βασικό είναι να υπάρξουν, υπάρξει ένα κοινό όρομα και νομίζω ότι προκύπτει ο κύριος Μπέρμαν κοίταξε και το σχέδιο έκθεσης του κύριου Μπροκ και τις προτινόμενες τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν. Η πρώτη του αντίδραση ήταν ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων. Σχεδόν όλες οι προτινόμενες τροπολογίες της ΑΦΕΤ αναφέρονται κυρίως και, αναφέρονται και στο σχέδιο γνωμοδότησης του Μπέρμαν. Μην πω την λέξη προς λέξη. στην γνωμοδότηση ΔΕΒΕ κάποιες τροπολογίες θέλουν να εισαγάγουν τις ε, εξή αλλαγέ στην πρόταση της Κομισιόν. Ε, έξι είναι τα βασικά σημεία. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στι αποφάσεις για τον προγραμματισμό και τις ε, αποφάσεις για την εφαρμογή. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα με την ΑΦΕΤ και ο Τάις και ο Χέλμαν Μπροκ συμφωνούν με τους προσανατολισμούς που έλαβαν από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η Κομισιόν και, το και την Κομισιόν και το Συμβούλιο, οτιδήποτε δεν είναι το νομοθετικό κείμενο θεωρείται εφαρμοστικό και εμπίπτει στους κοινού εφαρμοστικούς κανόνες ή εκτελεστικούς κανόνες. Για το Κοινοβούλιο όμως, διάφορες στρατηγικές ε, προγραμματικές αποφάσεις είναι σαφώς πολιτικές και θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει εντοπίσει αυτά τα στοιχεία ήδη το 2010. Οι ε, προτεραιότητες, ε, η επιλογή των προτεραιοτήτων και τα ποσά για το κάθε πρόγραμμα επίσης αναφέρονται. Οι τροπολογίες Μπροκ και Μπέρμαν υποβάλλονται για να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή. Και οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό να ενταχθούν στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης, όπως προβλέπει το άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μία σειρά από τροπολογίες που υπάρχουν για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το DCI ε, προϋποθέτουν ε, ότι Μιλάμε για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και ότι πρέπει να υπάρχει με βάση την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια επιλεξιμότητα. Ε, μπορεί εδώ πέρα να υπάρχει κάτι, ε, ειδικά στο ε, CIR, που, δεν έχει να, που είναι άσχετο με τα υπόλοιπα μέσα. Επίσης, σε μια δεύτερη σειρά τροπολογιών, ο Μπέρμαν μιλάει ε, για τη δυνατότητα να υπάρξουν αποτέλεσματα ε, από δράσεις ε, επί διαφόρων μέσων. Θέλουμε η Κομισιόν να μας λέει ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό μας οδηγεί ε, και στην εισαγωγή μιας ενδιάμεσης έκθεσης με τη δυνατότητα προσαρμογής και διόρθωσης της νομοθεσίας. Και επίσης θέλουμε κάποιες ημερομηνίε ε, για το δημοσιονομικό μέσο. η ε, ΑΘΕΤ και η ΔΕΒΕ συμφωνούν επ' αυτού. Τέταρτο σημείο. Κάποιες τροπολογίες θέλουν να περιορίσουν τις τις εξουσίες που θέλει να κρατήσει η Κομισιόν για τον εαυτό της. Ο Τας Μπέρμαν αναγνωρίζει την ανάγκη για ευελιξία και τη δυνατότητα που έχει η Κομισιόν να προσαρμόσει τα χρηματοδοτικά προγράμματα με βάση τις ε, γοργά ε, εξελισσόμενες ε, πραγματικότητες στην περίοδο 2014-2020. Αλλά θέλουμε να κρατήσουμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη δυνατότητα ε, μιας κάποιας έτσι προβλεψιμότητας στη χρήση δημοσίων κονδυλίων. Πέμπτον, μία σειρά τροπολογιών αφορούν τα άρθρα για τις δημόσιες προμήθειες ε, και την αποσύνδεση της βοήθειας. Η προτάση της Κομισιόν ε, κρατάει τις διατάξεις του σημερινού ε, μέσου αναπτυξιακής βοήθειας για την αποδέσμευση της βοήθειας. Υπάρχει μόνο μία αμφίσιμη πρόταση στο κείμενο της Προεδρίας, μία προβληματική πρόταση που αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι μέλη του G20 που δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαγωνισμούς που τρομολογούνται με βάση το DCI ε, και ε, το μέσο εταιρική σχέσης. Ο Μπέρμαν ήρθε σε επαφή με τον ΟΣΑ που το επιβεβαιώνει αυτή την ανάλυση ότι αυτό αντιβαίνει στις ε, κατευθυντήριες γραμμές της ε, αποδέσμες της βοήθειας υπό τον DCI. Δεν είναι αποδεκτό το να αποκλείσουμε κάποιες από τις αντισώμενες χώρες, γιατί θα έρθουμε σε αντίφαση με τις ίδιες τις πολιτικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δηλαδή θα αποδεσμεύσουν τη βοήθεια στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δέσμευση που την έχουμε επαναλάβει ε, σε υψηλό επίπεδο για την αποτελεσματικότητα της ε, βοήθειας πέρυσι. Τέλος. Μέσω της δουλειάς του που έκανε για το CIR και το DCI, μία από τις βασικές ανησυχίες ήταν να κρατήσουμε στις νομοθετικές προτάσεις τα κέρδη που πετύχαμε έξι χρόνια πριν όταν διαπραγματευτήκαμε το δημοσιονομικό α, μέσο που ισχύει αυτή τη στιγμή. Το DCI που ισχύει αυτή τη στιγμή έχει πολλές λεπτομέρειες και σε πολλά από αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή συζητάμε ούτω ώστε να τα προσαρμόσουμε Μιλάμε τώρα για μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί πριν από έξι χρόνια μεταξύ της Κομισιόν και του Συμβουλίου α, για το DCI. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτή τη συμφωνία. Το κατόφλι για να ξεκινήσει μια διαδικασία είναι πολύ ψηλό με βάση τα σημερινά δεδομένα. από τα 10 εκατομμύρια που είναι σήμερα έχει φτάσει στα 30. Αυτό είναι υπερβολικά ψηλό κατόφλι. Στον νέο κανονισμό μπορεί να φύγει αυτή η προϋπόθεση. Ε, ο Μπέρμαν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προϋπόθεση στο CIR. Στη Διαχειριστική Επιτροπή επίσης, όταν το EIB εμπλέκεται, ε, θα πρέπει να γίνονται οι διαβουλεύσεις. Ο Μπέργκμαν είπε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά που έχουμε ήδη στο DCI, στο μέσο δηλαδή αναπτυξιακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ο κ. Σαραζά και διάφοροι. Ευχαριστώ και χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί πριν τη συνεδρίαση, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε λεπτομερή σχόλια ε, κατόπιν εγκρίσεως των υπηρεσιών. Θα έρθουμε σε επαφή με τον εισηγητή για πιο εμπεριστατωμένε συζητήσει. Καλωσορίζουμε το σχέδιο τη γνωμοδότηση και διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι ουσιαστικά υποστηρίζει ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μικροδιαχείριση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική αρχή. Αυτό αναφέρεται ε, στη γνωμοδότηση, διατηρεί τα μέσα ευελιξίες και στους μηχανισμούς για την εξωτερική δράση για να μην γίνουν ουσιαστικέ αλλαγέ στα κατόφλια και στα όρια de για να υιοθετηθεί η διαδικασία εξέταση. Γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης και εξορθολογισμού πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξωτερικές δράσεις μας και φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να σταλεί ένα ε, ουσιαστικό μήνυμα στον ίδιο τον κανονισμό για αυτή την προσπάθεια ακριβώς απλούστευσης και θα θέλαμε να διατηρηθεί το άρθρο 1, ε, εδάφιο 3 διότι η τροπολογία 17 ζητεί να απαλληφθεί και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τις πιο ευέλικτες διαδικασίες ή τις πιο απλές τι πιο ευέλικτε. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να διατηρηθεί και όχι να διαγραφεί. Ενδιαφέρει πολύ του ενεχομένου. Η κατεξουσιοδότηση πράξη ε, ε, είναι μεν γενική εφαρμογή και ε, στα εκτός αν υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να βρούμε κάποια μέτρα για περισσότερη ευελιξία και καλύτερη υποπτία. Ε, των ε, προγραμμάτων. Στο προγραμματικό ε, έγγραφο πρόκειται για προγραμματισμό και όχι για την εφαρμογή. Δεν κα... λείπτεται από το CIR στο σύλλογό του. Υπάρχουν επιμέρους κανονισμοί που είναι ακόμα στο στάδιο του προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πράξεις κάτι εξουδότηση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξασφαλίσει συνέργειες και ε, συμπλήρωση μεταξύ του Μηχανισμού εξωτερική Δράσης και ε, Είναι όμως προσεκτική στην προσέγγιση της για να μην ε, ενταχθούν άκαμπτοι μηχανισμοί που θα ήταν αντιπαραγωγικοί καθώς είναι μεταβαλλόμενο το περιβάλλον. Εμεί θέλουμε να έχουν προβολή και να γίνονται ορατέ οι εξωτερικές μας δράσεις και ε, να συνεργαζόμαστε καλά με τους ε, εταίρους που εφαρμόζουν ε, επιτόπου αυτά τα προγράμματα, πράγμα που έτσι και γίνεται ήδη. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμίζει ότι μπορεί να συμφωνεί επί της ουσίας ε, της διατάξης που προτείνει ο εισηγητής, του σχέδιο της νομοδότησης, αλλά αυτές οι πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται ήδη ή θα συμπεριληφθούν ε, στις εφαρμοστικές διατάξεις ε, μετά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ξέρετε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσει αυτό το θέμα, είναι στον τριμερή διάλογο. Και γι' αυτό δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να επαναληφθούν και σε αυτή την ε, γνωμοδότηση τα όσα ισχύουν και παρακαλούμε η τροπολογία 37 να μην εγκριθεί. Υποστηρικτικά μέτρα τώρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είτε συμπεριλαμβάνονται ήδη στα προγράμματα δράσης, άρα ε, στην ίδια διαδικασία ε, επιτροπολογίας ή ε, δεν χρειάζονται καθόλου υποστήριξη ή ε, ε, οικονομική ή άλλες φορές μπορεί να χρειαστεί να εγκριθούν ξεχωριστά από τα προγράμματα δράσης. Ας πούμε οριζόντιες αξιολογήσεις ή ιστορικός οικονομικός έλεγχος. Γι' αυτό το άρθρο 3, εδάφιο 3 του CIR θα πρέπει να διατηρηθεί για να υπάρχει μια βάση ακριβώς για τα ανεξάρτητα αυτά μέτρα και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακαλούσε να αποσυρθεί η τροπολογία 33 του σχεδίου γνωμοδότηση. Ό,τι αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας, έχουμε ε, ήδη δεσμευτεί να βελτιώσουμε τη βοήθεια και να ε, βελτιώσουμε την ποιότητα, τη συνέπεια και τη διαφάνεια ε, ως προς τις αναφορές για το καθεστώς βοήθειας που χορηγείται. Παρόλο που επίσημη βοήθεια εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς εκτός του κανονισμού αυτού το CIR προσπαθεί να απλουστεύσει τους κανόνες και να εφαρμόζονται παντού σε όλα τα μέσα και ε, να διευρύνει ε, περαιτέρω ε, τους κανόνες επιλεξιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις σχετικές τροπολογίες που θέλουν ε, να διευρυνθούν αυτά ε, τα μέτρα σε όλες τις χώρες ε, του ΩΣΑ. Και επίσης πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με την εφαρμογή αυτών των μέτρων χώρες G20. Δεν αντιτίθεται η πρόταση CIR σε σχέση με αναπτυσσόμενες χώρες ή ε, χώρες που αναπτύσσονται με ταχύς ρυθμούς. Σε αναδυόμενες ε, οικονομίες μπορούν να επιβληθούν κάποιοι κανόνες του G20 που αφορούν τις αναπτυγμένες οικονομίες. Εκεί αλλάζουν οι κανόνες ανάθεσης σε διαγωνισμούς στις κρατικές προμήθειες ε, ε, δεδομένης της σημασίας της χώρας και της οικονομίας ε, στα διεθνή τεκτενόμενα. Υπάρχουν όμως χώρες που χρηματοδοτούν σε αυτή την περίπτωση της δράσης. Ε, και τελικά από, από χώρες αποδέκτες γίνονται χώρες δωρητές. Ευχαριστώ πολύ. Alors, euh, si vous permettez, je voudrais quand même Λοιπόν, εάν επιτρέπετε θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, η κατεξουσιοδότηση πράξης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που θα ήθελε η κατεξουσιοδότηση πράκτης, πράκτης πράξεις να προβλέπονται στον προγραμματισμό. Και δίνω το λόγο στον ε, κύριο Νόιζερ. Ευχαριστώ, κυρία Στρίφλερ. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι συζητάμε εδώ ένα πολύ τεχνικό θέμα. Mm-hmm. Αλλά οι ε, επιπτώσεις της αναπτυξιακής πολιτικής θα είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τις χώρες που αποκλείονται από το G20, ε, ε, πρέπει να γίνει μία προσπάθεια για να περιληφθούν αλλά πιστεύω ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τις κατευθυντήριες γραμμές του DIC. Ε, εξού και πιστεύουμε σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες μας έχουν δοθεί ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στο DIC μετά τις θερινές διακοπές και πιστεύω ότι το DIC είναι ο χώρος όπου θα πρέπει να αποφασιστούν οποιασδήποτε αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε μετά τις θερινές διακοπές και θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα του G20. Ευχαριστώ. Προτείνω ότι ε, προθεσμία για τις τροπολογίες είναι για αύριο το πρωί και περνάμε στο επόμενο θέμα. Περιμένουμε βέβαια την γνωμοδότηση ε, του Υπουργού, αλλά επειδή είμαστε λίγο μπροστά στο πρόγραμμά μας, προτείνω να κάνουμε ε, μία διακοπή 5 με 7 λεπτών. Euh, Είναι, ε, ε, ε, έρχονται οι υπεύθυνοι, άρα πέντε λεπτά νομίζω θα επαρκέσουν. Merci. Καθίστε παρακαλώ. Και να χαμηλώσετε λίγο τις ομιλίες σας, τη φωνή σας. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας για δεύτερη φορά τον κύριο Κρίστιαν Φρίσμπαχ, Δανό Υπουργό της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη. Στην προηγούμενη επίσκεψή σας, κύριε Υπουργέ, τον Φεβρουάριο, είπατε ότι είσαστε στη διάθεσή μας, θα θέλατε να επανέλθετε εδώ πριν από το τέλος της ε, Δανέζικης Προεδρίας για να τα ξαναπούμε. Μεγάλη χαρά λοιπόν σας ξαναβλέπουμε σε αυτή τη δεύτερη επίσκεψή σας. Ο σκοπός της ε, σημερινής σας επίσκεψης είναι να μας παρουσιάσετε στην Επιτροπή μας τα αποτελέσματα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ε, Εξωτερικών Υποθέσεων ε, της 14ης Μαΐου που ασχολήθηκε με την συνεργασία για την ανάπτυξη. Από ό,τι καταλάβαμε, ε, η κυρία Άστον, που είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο όνομα αυτής μας κάνετε αυτή την έκθεση. Σε αυτή τη συνεδρία συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα για την Επιτροπή μας, καθώς και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανάπτυξη. Οι Υπουργοί συζήτησαν την ανακοίνωση του Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για το πρόγραμμα για την αλλαγή και το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το μέλλον και η, της πολιτικής αυτής και η δημοσιονομική υποστήριξη, καθώς και της διετούς έκθεσης για την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Παρακαλώ μην μιλάτε, δεν μπορώ παράλληλα να σας ακούω. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία, ε, ετοιμαζόμαστε, για τα οποία ετοιμαζόμαστε να υιοθετήσουμε συστάσεις στο Κοινοβούλιο. Ο συνάδελφος Σάρλ Γκέρενς ε, μόλις τελειώσε την έκθεσή του για το πρόγραμμα για την ανάπτυξη ε, και την δημοσιονομική βοήθεια και η συναδελφός μας Μπρίγκιτ ε, Σνάιμπερ Γιάστραμ ολοκληρώνει την έκθεσή της για την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Θα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας ε, επί των εργασιών του Συμβουλίου. Έχετε περίπου το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και εκπροσωπώ την ύπατη ε, εκπρόσωπο την κυρία Άστον και, σας, και θα σας ενημερώσω για το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου στις Βρυξέλλες. Όπως ε, ανακοινώθηκε από τη Βαρόνια Άστον, θα κάνουμε ε, μόνιμες επαφές, θα έχουμε μόνιμες επαφές με την Επιτροπή Ανάπτυξης, όπως κάνουμε και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για ενημέρωση. Προσωπικά τώρα χαίρομαι που ξαναέρχομαι εδώ, γιατί βρίσκω ότι η συζήτηση τελευταία φορά είχε πολλές αιχμές, πολλές προκλήσεις, αλλά και ήταν πολύ χρήσιμη. Και μου άρεσε πολύ η συζήτηση που είχαμε μερικούς από εσά που συμμετείχατε σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Όσλο. Μπορώ να σας πω ότι το Συμβούλιο Υπουργών είχε καλά αποτελέσματα. Καλή η συμμετοχή των Υπουργών, 15 από τις 27 συμμετείχαν, Τέσσερις ώρες συζητήσαμε, κάναμε σοβαρές πολιτικές συζητήσεις και λάβαμε και σοβαρές αποφάσεις. Ε, τους τελευταίους έξι μήνες υπάρχει σημαντική πρόοδος για σημαντικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη. Και αυτό το σημείωσε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, εκπρόσωπος, αλλά και πολλά κράτη-μέλη. Διάφορα μεγάλα θέματα, η ατζέντα για την αλλαγή, το πρόγραμμα διαδράση για την αλλαγή, το, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μιανμάρ, ε, το Ρίο 20, ε, επίσης, ε, τα συμπεράσματα για την ε, επιστηστική ασφάλεια στο κέρας της Αφρικής και γενικά η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Θα ξεκινήσουμε την ατζέντα για την αλλαγή. Οι ΥΠΑΤΙ εκπρόσωπος και οι Υπουργοί καλωσορίζουν τη σημαντική πρόοδο που έγινε από τη συζήτηση του Νοεμβρίου και μετά. Και υπάρχουν τρεις τομείς πρόοδου. Καταρχάς, συμφωνία ούτω ώστε η αναπτυξιακή πολιτική να βασιστεί σε, σε δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα από τη μία και ε, ανάπτυξη με συμμετοχή όλων από την άλλη. Αυτοί είναι δύο βασικοί πυλώνες που θα αποτελέσουν ε, ε, τη βάση της αναπτυξιακής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, δέσμευση. Ε, η, βοήθεια να εστιαθεί σε λιγότερους τομείς και σε πιο φτωχές, ε, στις πιο φτωχές χώρες, ώστε να μειωθεί η φτώχεια. Επίσης, θα πρέπει να βλέπουμε πώς θα πηγαίνουν στην ε, δημοκρατία στα ανθρώπινα δικαιώματα οι εταίροι μα. ειδικά όταν μιλάμε για δημοσιονομική συγγνώμη στήριξη. Υιοθετήθησαμε συμπεράσματα για την ατζέντα για την αλλαγή και θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλεύουν ε, πιο αποτελεσματικά και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Επίση, θα υπάρξει η αρχή τη διαφοροποίηση και η βοήθεια θα εστιάζεται και θα δίνεται στις πιο φτωχές χώρες. Θα πρέπει να έχουμε... Ορισμένοι μίλησαν για αλλαγέ στη Λατινική Αμερική, ορισμένοι ζήτησαν να σταλεί ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα γενικά στι ε, χώρε που βοηθούνται. Πολλοί υπουργοί ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής ε, και στην αναθεώρηση που θα κάνουμε της πολιτικής μας και στην ε, συζήτηση με άλλους εταίρους και οι υπουργοί ε, καλωσόρισαν την υιοθέτηση των σχετικών συμπερασμάτων Συμβουλίου. Υπήρξαν πολλέ ε, παρεμβάσει ε, υπέρ του σημερινού προγραμματισμού, που θα είναι μια διαδικασία αναχώρα. Και τα κράτη-μέλη που, δεν που δεν είναι παρόντα επιτόπου, δεν δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να ενημερώνονται παρόλα αυτά για την πρόοδο. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι ευκαιρίε, ούτω ώστε να έχουμε κοινού προγραμματισμού στι χώρε, όπου υπάρχει ελπίδα, αλλά η πρόοδος δεν είναι σημαντική. Σε ορισμένε χώρε όπω την Αιθιοπία ε, υπήρξε συμφωνία για να εξηγήσουμε καλύτερα τα ωφέλη του κοινού ε, προγραμματισμού ε, και να τα εξηγήσουμε και στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων. Επίσης, όλα αυτά εξαρτώνται από την πρόοδο που υπάρχει από τις χώρες αυτές στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Αυτέ οι βασικέ αξίε θα πρέπει να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα και θα πρέπει να υπάρχει, ζητείτε να υπάρξει μεγαλύτερη αξιολόγηση. Ε, επίσης, συνεργασία ε, και συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το συζήτησαν πολλοί υπουργοί. Τώρα, οι στόχοι τη βοήθεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα στη σημερινή δημο, δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση. Οι τάσει του ΩΣΑ δείχνουν μια μεικτή εικόνα εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο, παραμένουμε, αλλά όλο και μικρότερα είναι τα ποσά που δίνει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθειά μας. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έχει μειωθεί σχετικά, οριακά μάλιστα, από το, το 2010 και 2011 στα 53,1 δισεκατομμύρια ευρώ. και από το 0,44 του ΑΕΠ μας έχει φτάσει τώρα στο 0,42%. Ε, για να πετύχουμε τους στόχους το 2015 όμως θα πρέπει να διπλασιαστεί η βοήθεια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια βασική ισορροπία στα πολιτικά μηνύματα που θα δώσουμε. Τα κράτη-μέλη τα οποία ε, ξεπερνούν το 0,7 του ΑΕΠ τους ε, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους, όπως και εκείνη που η βοήθειά τους το 2011 ήταν πάνω από τους στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010. Ε, κάποια κράτη-μέλη μίγασαν για, την, για τη λιτότητα, την δημοσιονομική πειθαρχία και την οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά τόνισαν την πολιτική ευθύνη που έχουν και την προσπάθεια κινητοποίηση δημόσια ε, της κοινή γνώμης για εστιασμένες συλλογικέ προσπάθειες. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την διάσκεψη του Ρίο Plus 20 για να εφαρμόσουμε του τους στόχους και να αρχίσουμε μια διαδικασία προβληματισμού για το ρόλο τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μετά το 2015. Η ύπατη εκπρόσωπος τόνισε ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια εξυπηρετεί και τα δικά μα συμφέροντα και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια ούτω ώστε να το κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, να κατανοήσουν τη σημασία τη βοήθεια αυτή και τα αποτελέσματα μα βοήθησαν να πετύχουμε. Και ζήτησε από όλου του υπουργού να αυξήσουν τι προσπάθειε του για να υλοποιήσουν του στόχου τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Στα συμπεράσματα, ε, όλα τα κράτη-μέλη ε, είπαν ότι θα αυξήσουν μέχρι το 2015 την αναπτυξιακή του βοήθεια στο 0,7% του ΕΠ και ξανατόνισαν τις, ε, τη δέσμευση ε, των εθνικών και συλλογικών στόχων. Δεν θα σε εκπλήξει ότι η Μιανμάρ είναι πολύ σημαντικό θέμα μετά την επίσκεψη και της κυρίας Άστον αναφέρθηκε στη μοναδική διαδικασία που είναι εξελίξη και στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση ε, με κοινό προγραμματισμό, να βασιστούμε στις υπάρχουσες δομές βέβαια, αλλά να υπάρξει και μεγαλύτερος και πιο, πιο έντονος διάλογος και να υποστηρίξουμε την μεταβατική διαδικασία, να διατηρήσουμε το διάλογο με την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις αυτής, ούτως ώστε να υπάρξει και βιώσιμη ειρήνη και με τις διάφορες κοινότητες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να παίξει συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημαντικό ρόλο και ο Επίτροπος ε, υποστήριξε την ε, παρέμβαση της κ. για τις οικονομικές δεσμεύσεις ε, του 2012, 100 εκατομμύρια ευρώ και το 2013 50 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει δημιουργία δυναμικού. Θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκός συντονισμός, το υποστήριξαν όλοι αυτό, και μία ε, προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα και στην, σε μια αποτελεσματική χορήγηση της βοήθειας. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Επίσης, μίλησε ότι θα πρέπει να υποστήριξουμε τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Κάποια κρατημένα αναφέρθηκαν στην ανάγκη να βασιστούμε από τη δική μας εμπειρία, τη μεταβατική εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε σχετική εμπειρία στον τομέα της συμφιλίωσης. Ε, στη συζήτηση επίση είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμε δεσμεύσει, μια συντονισμένη δράση, συνένεση, ούτω ώστε να δούμε τι δυναμικό υπάρχει για κοινό προγραμματισμό με την Βυρμανία Μιανμάρ. Ε, επίσης, Ρίο πλάς 20. Είπατε εκπρόσωποι, πως και πολλοί υπουργοί είπαν ε, ότι πρέπει να συζητήσουμε ε, και την σημασία της ανάπτυξης στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Επίτροπος Ποτότνεκ υπενθύμησε τις διάφορες πτυχές της ατζέντα του Ρίο και τις θέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις και υπήρχε βρία συμφωνία των κρατών μελών ότι η διάσκεψη του Ρίο θα πρέπει να θεωρηθεί και αναπτυξιακή διάσκεψη. Θα πρέπει να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνικό πυλώνα και περιβαλλοντικό πυλώνα, τρει πυλώνε δηλαδή, που θα τη στηρίζουν. Επίση, η συζήτηση έδειξε ότι η πράσινη οικονομία ε, έχει και μια κοινωνική διάσταση και συμπεριλαμβάνει την επιστημιστική ασφάλεια, την υγεία κτλ και μια μετάβαση προς την πράσινη οικονομία είναι πρόκληση για όλες τις χώρες και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει όμως και σημαντικά ωφέλη για όλες τις χώρες. Ε, πολλά κράτη-μέλη ανέφεραν την, ε, τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης ως πιθανό ε, αποτέλεσμα της διάσκεψης ΡΙΟ που θα πρέπει να συντονιστεί με τη διαδικασία αναθεώρησης των στόχων της χιλιατίας που είναι εξελίξη και να μην ε, προχωρήσουμε σε δύο παράλληλες ατραπούς. Δεν πρέπει τα στόχους της ηλιετίας και του στόχου του ουρίου να τους βλέπουμε χωριστά. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι στόχοι της ανάπτυξης είναι τελείως διαφορετικοί και δεν θα πρέπει εμείς ε, να δημιουργήσουμε προσκόμματα στη διαδικασία ε, υλοποίησης των αποτελεσμάτων και επιτευχτών στόχων. είδαμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε και χωριστό συμβούλιο που θα ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ορισμένοι είπαν ότι υπάρχουν αρκετέ ήδη δομέ και φορεί, παραδείγματο χάρη η ΕΟΚΕ, ε, και θα πρέπει να του λάβουμε υπόψη μα, ειδικά αν θέλουμε να προχωρήσουμε και την ιδέα τη καινοτόμου χρηματοδότηση. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν. Υπήρξαν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα διάφορα. Ε, ο Επίτροπος Πίμπαλξ ενημέρωσε για τα συμβάσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της αντοχής στις επιστημικές κρίσεις στο κέρος της Αφρικής. Υιοθετήθηκε την ίδια ημέρα αυτό το συμπέρασμα και τονίζεται η σημασία δεσμών μεταξύ της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για να υπάρξει αυτή η αντίσταση στις κρίσεις. Ο Επίτροπος Πίμπαρξ μας ενημέρωσε για την ε, πρωτοβουλία του G8 για τη νέα πρωτοβουλία για την επιστημική ασφάλιση που αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο του G8 για να υπάρξουν ιδιωτικές επενδύσεις στη Αιθιοπία Μοζαμβίκη, Αιθιοπία, ε, Γινέα Μπισάου, έξι αφρικανικές χώρες ε, ούτως ώστε μέσα 10 χρόνια ε, να βοηθήσουμε 50 εκατομμύρια Αφρικανούς. Στις 11 Ιουλίου ε, στο Λονδίνο ε, θα συζητηθεί το θέμα του οικογενειακού προγραμματισμού και θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε κοινούς προγραμματισμούς με διάφορες χώρες, τρίτες χώρες εταίρους. Αυτά είναι όλα τα θέματα που καλύφθηκαν. Τώρα είμαι έτοιμος για να το συζητήσουμε, να ακούσω τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας. Και σε ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση των πεπραγμένων του Συμβουλίου. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και σας προσωπικά και τη Δανική Προεδρία για την κοινοβουλευτική συνέλευση με τις χώρες ΑΚΕ την περασμένη εβδομάδα στη Δανία και άκουσα από συμμετέχοντες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕΝ να εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση. Χάρηκαν πάρα πολύ για το υψηλό πολιτικό επίπεδο όσο και για την ουσία. Ήρθε η Πρωθυπουργό της Δανίας, Τρει επίτροποι. Ήταν πολύ υψηλού επίπεδου η πολιτική συνάντηση αυτή. Και αυτό το εκτίμησαν. Στο παρελθόν ήταν χαμηλότερο το επίπεδο των πολιτικών ε, αξιωματούχων. Αφήστε δε και τη δανεική φιλοξενία που δεν χρειάζεται να πω τίποτα γι' αυτή. Ε, ευχαριστώ πολύ Υπουργέ και παρακαλώ διαβιβάστε τα δέοντα και στην Πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούσαμε σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ε, συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. PCD είναι τα αρχικά στα αγγλικά. Ακούσαμε και το βλέπουμε και στα συμπεράσματα της Προεδρίας ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε πέντε προτεραιότητες. Εμπόριο, χρηματοδότηση, ε, κλιματική αλλαγή, ε, επιστηστική ασφάλεια και μετανάστευση. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η συζήτηση ε, ήταν περιορισμένη στις πέντε προτεραιότητες ή ευρύτερη. Γιατί ε, γνωρίζουμε ότι τα θεσμικά όργανα εργάζονται για τις μεταρρυθμίσεις ε, και αυτό θα επηρεάσει και την ανάπτυξη. Εδώ αναφέρομαι και στην κοινή γεωργική πολιτική και στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν καθόλου και αν ναι, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τελικά στις προτεραιότητες, στις πέντε θεματικές ενότητες. Καλωσορίζω αυτή τη ε, ανακοίνωση ότι στο μέλλον, στις συνεδριάσεις των Υπουργών ε, εξωτερικών και γενικών υποθέσεων θα βρει μεγαλύτερο χώρο το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Τρεις-τρεις, ο κύριος Κοτνορτές Λάστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, χαρά μας που σας βλέπουμε εδώ ενώπιόν μας. Το είπα και στην αρχή της Προεδρίας όταν ήρθατε και πραγματικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενέστατα αυτά τα θέματα μαζί σας. Χαίρομαι που ήρθατε για να μας αναφέρετε και στο τέλος της ε, Δανικής Προεδρίας. Και σας ευχαριστώ πάντα για τη στάση που για τη ρήτη απέναντι στην Επιτροπή μας. Δύο ερωτήσει αρκετά συγκεκριμένες, γιατί θα σας ρωτήσω και άλλοι συνάδελφοι γενικότερα. Το ένα, οι στόχοι της ε, χιλιετίας, θυμάστε για το 2015, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό και μας απασχολεί και μας στην Επιτροπή μας. Τι γίνεται μετά το 2015 με τους στόχους αυτούς και τι γίνεται και μέχρι το 2015. Το συζητήσατε σε αυτή τη συνεδρίαση υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα πορευθούμε μέχρι το 2015. Ε, πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Κάποια στιγμή αναφερθήκατε στις λεγόμενες ε, συνεργασίες τριγωνικού τύπου, συνεργασία χωρών του Νότου με άλλες χώρες του Νότου κτλ. Και προσθέτω και μια τρίτη ερώτηση για το Σαχέλ. Η Επίτροπος Γεωργίευα πριν από λίγες εβδομάδες είχε έρθει εδώ και μας είπε ότι ανησυχεί, όπως και εμείς άλλωστε στην Επιτροπή μας, σε σχέση με την κατάσταση στο Σαχέλ. Μας είπε ότι το 50% της ανθρωπιστικής βοήθειας πηγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Η μισή βοήθεια είναι της Ένωσης που φτάνει στο Σαχέλ. Αυτή η βοήθεια νομίζω ότι θα πρέπει να αυξηθεί, είναι πολύ σημαντικό να είναι στο ύψο των περιστάσεων ε, η Ένωση και αν δεν αυξηθεί ή ποτέ να μην μειωθεί, να μην σηκώσουμε ποτέ τα χέρια ψηλά στην ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στο Σαχέλ που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θα πρέπει να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν μου επιτρέπετε, η πρόεδρο, τέταρτη ερώτηση από τι δύο που είχα αρχικά, με τα πέντε βασικά σημεία τη προτεραιότητα συνδέεται και μία από αυτέ είναι η ασφάλεια. Θα ήθελα να ρωτήσω, σας απασχόλησε αυτό, πώς θα συνδέσετε την ασφάλεια με τη συνεργασία συγκεκριμένα, όχι γενικά ασφάλεια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, je passe la parole... Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκέρενς. Και μετά απαντήσεις σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Και έχω άλλους τρεις μετά. Παρακαλώ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν διαβάσουμε τα συμπεράσματα ενός Συμβουλίου, λέμε ότι τα καταλαβαίνουμε καλύτερα αν ε, έχουμε συμβάλει στη σύνταξη των συμπερασμάτων. Αλλά αυτά τα συμπεράσματα είναι αρκετά σαφή και μπορούμε να πούμε ότι έξι τον κόπο να γίνει αυτό το Συμβούλιο διότι Άκουσα ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε και ε, στην εισαγωγή ε, του αναφέρθηκε σε 15 υπουργούς και ακόμη περισσότερους ε, υφυπουργούς. Πρώτη φορά ακούμε κάτι τέτοιο ε, και μέχρι τώρα ε, ποτέ δεν είχαμε δει να συμμετάσχουν 15 υπουργοί και είναι η πρώτη φορά που κάποιος ε, μπορεί να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα και το χαιρετίζω διότι αντιλαμβάνομαι ότι η εργασία την οποία κάναμε υπέρ μιας καλύτερης λειτουργίας των θεσμικών οργάνων δεν πήγε στράφη και χαιρετίζω την δραστηριότητά σας σαν Υπουργό και τον τρόπο με τον οποίο σας εμπιστεύονται οι ευρωπαϊκές αρχές για να, μπορέσουν να, για να μπορέσετε να παρουσιάσετε εδώ, εδώ τα συμπεράσματά σας και έχω εδώ δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω για το Ρίο 20 ε, υπάρχουν συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και θα μπορούσαν ενδεχομένως να θίξουν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ποιο τομέα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία μας παρουσιάσατε να γίνουν πραγματικότητα. Και δεύτερον, ένα θέμα το οποίο παρουσιάστηκε πολύ ανώδυνα είναι το σημείο 16 ε, που επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά προέβη στα σχόλια για τη διαφοροποίηση της ενισχύσεως. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί στην Επιτροπή μας αλλά με τα χαράς διαπιστώνω ότι το Συμβούλιο μπόρεσε να συμφωνήσει επί μιας κοινής γραμμής σε αυτό το θέμα γραμμή την οποία ε, ε, συμμερίζομαι και ιδίως όσον αφορά το phasing out αλλά η αρχή νομίζω ότι έχει γίνει θετικά αποδεκτή από το Συμβούλιο και αυτό είναι ευχάριστο νέο, συμφωνεί με τη λογική και ε, έτσι πρέπει να κινούμαστε. Ερώτηση. Το phasing out αυτό συζητήθηκε πιο λεπτομερώς διότι στην περίπτωση αυτή θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες ε, σχετικά με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Εάν κάτι παραλείψω, παρακαλώ να, ε, μου το ξαναζητήσετε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω για ε, όσους συμμετείχαν στη Δανία στην συνεδρίαση όπου έγινε κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή. Χάρηκα από πολύ διότι οι συζητήσεις οι οποίες διεξήχθησαν και οι δραστηριότητες πέραν του επισήμου προγράμματος ήταν ευχάριστες και υπήρξαν γεύματα ε, με τους πολίτες, με την κοινωνία των πολιτών, ένα αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ε, της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ευρωβουλευτών και ε, βουλευτών και ε, τα θέματα αυτά τα οποία είναι ευαίσθητα τα θίξαμε και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Βέβαια, ε, όσον αφορά την συνεκτική ανάπτυξη ε, συμφωνήσαμε, αναφερόμαστε σε πέντε τομείς ε, η ασφάλεια ήταν το ένα θέμα μία επιχειρησιακή προσέγγιση ήταν το άλλο και μία στενότερη συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών ήταν επίσης χρήσιμα και αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν πιο εκ του με γειτονικές χώρες κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική με χώρες εταίρους ε, μέσω των ε, εκπροσωπήσεών τους και στο μέλλον. Βέβαια, η κοινή πολιτική αλληλείας και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει επίσης ε, να ισχύσουν και δεν μπορούν να γίνουν ε, χωρίς να λάβει κανείς ε, υπόψη τις παρενέργειες ορισμένων θεμάτων και όσον αφορά την πολιτική αλληλεία θα πρέπει κανείς να τονίσει και την διάσταση τη βασική που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν κανείς ε, ε, εξετάζει τις αρχές που την, ε, τι, οι οποίες διέπουν αυτή την πολιτική και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και μία οικονομική συζήτηση σχετικά με τον κύριο Λάστρα. Η διαδικασία σχετικά με τους στόχους της χιλιετηρίας ε, ξεκινά από το 2013 και ε, έχει καταρτιστεί ένα, μια ομάδα υψηλού επίπεδου που θα παρακολουθεί τα θέματα μετά από τη διάσκεψη κορυφής και που στη συνέχεια θα μπορέσει να επηρεάσει και τις συζητήσεις μέχρι την αναθεώρηση των στόχων της χιλιετηρίδος. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα υπάρχει ένας στενός διάλογος επί του θέματος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που θα εξετάζει ε, τις ε, κοινές πολιτικές στα πλαίσια του ε, προγράμματος του 2015 και τονίσαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμους στόχους και στόχους της χιλιετηρίδας οι οποίοι δεν θα συγκλίνουν και είναι κάτι που θα πρέπει να συζητείτε από κοινού. Αυτή είναι η απόφαση η οποία συζητήθηκε και λήφθη αλλά σχετικά με τη συζήτηση μετά το 2015 θα ξεκινήσει ουσιαστικά μετά τη διάσκεψη κορυφής όπου θα υπάρξει ενημέρωση και θα εδρεωθεί η συμβουλευτική ομάδα ε, για να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία αναθεώρησης ε, των στόχων της χιλιατηρίδος ε, που προβλέπεται. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και προβλέπεται εις, ε, τα συμπεράσματα της ατζέντα για την αλλαγή και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από πολλά κράτη συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου έχουμε περιλάβει την συνεργασία με τους νότιους ε, εταίρους και για να μιλήσω για τους Δανούς έχουμε τώρα τριμερείς συμφωνίες με τη Βραζιλία, με την Νότια Αφρική, την Νότια Κορία, Κορέα ε, και άλλες χώρες και γίνονται προσπάθειες να καταρτιστούν τρεις, τριμερείς συνεργασίες, αναπτυξιακή συνεργασίας ε, με τρεις, μεταξύ τριών χωρών και ε, η, και η ε, Κίνα μας ζήτησε να ενημερώνεται για την ε, ατζέντα του Πουσάν και την έκβασή της διότι ενδέχεται και αυτοί να θελήσουν να εμπνευστούν και να οθηθούν από τις αρχές αυτές. Συμφωνώ μαζί σας σχετικά με την περιοχή του Σαχέλ. Πρόσφατα επισκέφτηκα την περιοχή και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ βασικός παίκτης όπως πολύ σωστά τονίσατε μέσα στα πλαίσια της ε, συνεκτικής ε, ε, στρατηγικής για το Σαχέλ που είχαμε πέρυσι κινητοποιήσει 150 εκατομμύρια ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει κινηθεί ενεργά ε, υπέρ της ε, ανθρωπιστικής βοηθείας. Είναι όμως ένα πολύ περίπλοκο θέμα όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα και είναι ανάγκη να υπάρξει μία καλύτερη προσέγγιση το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα για τον Βόρειο Νίγηρο όπου υπάρχουν δύο προγράμματα που πρέπει να συνυπάρξουν ε, και ε, βλέπουμε ότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζουν και πρέπει να προωθήσουμε αυτή την προοπτική ε, προβλέποντας και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενσωματώνοντας φορτώνοντας ε, αυτές τις πτυχές ε, στην βοήθεια προς το Σαχέλ. Όλα αυτά ουσιαστικά ε, όντως έχουν ληφθεί υπόψη και είδα ποια είναι η, πώς συνδυάζονται η κλιματολογική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση, και πόσο πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ε, κύριε Γκέρεν, σε ονόματι του Συμβουλίου βεβαίως ε, ε, θέλουμε να συναντηθούμε να διερευνήσουμε τα θέματα αυτά περαιτέρω και εγώ χαίρομαι προσωπικά που συμμετέχω σε αυτό τον διάλογο. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας για το Ρίο, θέλετε να δείτε πώς η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, προχωρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την διαπραγματευτική της θέση Πέραν αυτού όμως έχω διαπιστώσει στις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τι γίνεται στη Νέα Υόρκη ότι υπάρχει μία μετριασμένη αισιοδοξία ε, η οποία έχει εκφραστεί, η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει γίνει αντιληπτή ιδιαιτέρως όσον αφορά το κείμενο και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται να αναθεωρηθεί ή να προσαρμοστεί αλλά ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια έχουμε ε, δει τους βασικούς στόχους και σε ορισμένες ε, υποανάπτυξη χώρες υπήρξε ε, μία παρανόηση σε τομείς οι οποίοι δεν κατανοήθηκαν σωστά. Πιστεύω μάλιστα ότι αυτές οι παρανοήσεις διευκρινίστηκαν. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ε, αλλά να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και αν μιλάμε για θέματα σαν το νερό ή την ενέργεια, ή την διαχείριση των φυσικών πόρων δεν είναι ε, θέματα ε, μεμονωμένα αυτά αλλά είναι θέματα πολύπλοκα που έχουν σχέση με όλες τις πτυχές. Το νερό είναι σημαντικό ε, περιβαντολογικά αλλά συγχρόνως και από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε διάφορα θέματα τα οποία να διατυπωθούν πιο γενικά. Εξού και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος ελπίζω να προχωρήσει. Όσον αφορά τα θεσμικά θέματα, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις ε, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την, ε, την, ε, την δυνατότητα απολογισμού, σε ποιον θα πρέπει να αναφέρεται κανείς στο, στην Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση. Εγώ μιλώ σαν δανός βέβαια και πιστεύω ότι ε, ένα Συμβούλιο Βιωσιμότητος δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί σε μικρό επίπεδο, άρα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλη την αλυσίδα ανάληψης ευθυνών και πρέπει στην Αφρική να μπορέσουμε να προωθήσουμε διάφορα θέματα και ελπίζω ότι αυτό θα το δούμε και στο Ρίο. Διαφοροποίησης. Δηλαδή, μέχρι που θα μπορέσει κανείς να προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο ε, ε, ψηφίστηκε από το Συμβούλιο, η διαφοροποίηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε πίσω χώρες, διότι θα υπάρχουν διάφορα είδη συνεργασιών που θα προωθηθούν και θα υπάρξει ένα νέο είδος συνεργασίας που θα αναπτυχθεί με τις χώρες αυτές και θα υπάρξουν και θεματικά μέσα για χώρες όπου επηρεάζεται η συνεργασία. Δεν θα αφήσουμε δηλαδή ορισμένες χώρες πίσω, θα χρειαστεί να εκπονήσουμε νέους τρόπους συνεργασίας ε, που θα επηρεάσει και στο μέλλον ε, τον καταμερισμό της χρηματοδότησης χρηματοδότησης και θα υπάρξει και ε, μία σειρά χωρών με, όπου ε, η αναπτυξιακή βοήθεια θα εκπνεύσει και αυτό συζητιέται στο Συμβούλιο και από πλευράς εφαρμογής και από πλευράς διεκπαιρεώσεως. Αλλά θα δούμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς αυτό μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο ακόμη συζητείται στα πλαίσια των ε, διαφόρων εργαλείων και η εφαρμογή θα είναι ε, και ένα μέρος του διαλόγου με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Έχουμε άλλα τρία άτομα τώρα που ζητάνε το λόγο. Ο κύριος Μπέρμαν ο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας, Υπουργέ, για την παρουσίαση και τις απαντήσεις που απαντάνε και μέρη στις ερωτήσεις μου. Ε, θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα πράγματα για την Δυτική Αφρική. Μιλήσατε για τη Σαχέλ, μιλήσατε για την Κινέα Μπισάου, που δεν είναι τμήμα τη Σαχέλ. Υπάρχει μια μαζική αποσταθεροποίηση στην ε, Δυτική Αφρική, που είναι ανησυχητικό από στρατηγική άποψη για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε σταθερότητα στην περιοχή, χρειαζόμαστε κράτο δικαίου. Θέλουμε να υπάρχουν αποτελεσματικέ δομέ ούτως ώστε και οι σαλαφικές, ε, τα σαλαφικά κινήματα να, τα, να αντισταθούμε σε αυτά ε, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κτλ. Πώς βλέπετε την ανάγκη να επενδύσουμε πολύ και πολιτικά και υλικά για να εξασφαλίσουμε αυτή τη σταθεροποίηση στην περιοχή. Δεύτερη ερώτηση. Όχι δώσω για τη διαφοροποίηση, γιατί απαντήσατε σε αυτό αλλά για την έκθεση ομοτήμων της ΩΣΑ ΕΑΒ. Δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Έχει συζητηθεί και αν ναι, ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα. Βλέπω εδώ τον κύριο Ποπόφσκι, αλλά ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα, αν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Βεβαίω, ε, ήρθα λίγο καθυστερημένος, επειδή έμπλεξα σε κυκλοφοριακό από 0,44 ε, φτάσαμε στο 0,42 του ΑΕΠ στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ποια πρωτοβουλία μπορείτε να πάρετε ούτω ώστε να αντιστρέψετε αυτή την τάση που υπάρχει και ούτω ώστε η κοινή γνώμη ε, να συνταχθεί με την αντιστροφή αυτής της τάσης, να δεχθεί δηλαδή να αυξηθεί ακόμα το ποσοστό του ΑΕΠ που δίδεται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα επαναλάψω θα επαναλάβω ουσιαστικά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κάσμαρεκ σχετικά με τη συνεδρίαση και ισχύει και για την συνεδρίαση ε, της ε, Κοπενχάγης. Ήταν όντως τόσο καλή ώστε διότι η Ιδανική Προεδρία είχε προετοιμάσει τα πάντα πολύ ωραία, συμμετείχε και ο Δανός Πρωθυπουργό συναντώ τον Υπουργό τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα είναι μια τιμή για μένα και πιστεύω ότι η Προεδρία της Δανίας θα έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη σχετικά με την μέτρηση επιδόσεων των επομένων Προεδριών του Συμβουλίου. Εν ονόματι λοιπόν πολλών συναδελφών από τις χώρες ΑΚΕ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την αποτελεσματικότητα, τη φιλοξενία, την επιλογή των θεμάτων ότι η καλή συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο και οι ανανημόσιμες πηγές ενεργείας ήταν εξαιρετικά θέματα προς συζήτηση και οι εκδηλώσεις επίσης. Όσον αφορά την Agenda of Change θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ουσιαστικά υπολείπεται των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κατά τη γνώμη μου δεν, ε, ε, δεν υποδηλούν ότι θα καταλήξουμε σε μία ενιαία συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά μάλλον σε ένα σύστημα το οποίο θα περιοριστεί σε μερικές πιλωτικές χώρες ενώ χρειάζεται καλύτερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, πιο στενίες διαβουλεύσεις γι' αυτό και με απογοητεύομαι που το Συμβούλιο δεν ακολούθησε και έμεινε πίσω από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικό με τις συνθήκες και τις, ε, ε, κοινές, τους κοινούς προγραμματισμούς. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορούν να διευρυθούν για να επιτρέψουν μια καλύτερη συνεργασία με τις υποανάπτυξης χώρες. Κυρία Κρατή. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Χαιρετίζω όλα αυτά που κάνατε, εσείς προσωπικά και η Δανέζικη Προεδρία όλη αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τους στόχους της ε, χιλιετίας, αλλά ήδη το θίξατε και δώσατε κάποιες απαντήσεις. Να σας ρωτήσω τώρα, τι σημαίνει αυτή η αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας που είπατε. Οι λιγότεροι πόροι που έχουμε, δηλαδή εννοείται ότι θα πρέπει να ε, δοθούν σε λιγότερους ε, στόχους για την επίτευξη λιγότερων στόχων. Ή, όπως έχετε πει κατά επανάληψη, εννοείται την συζήτηση της μεταρρύθμισης των στόχων της χιλιετίας. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, είναι σαφές ότι το 2015 δεν θα έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι και ίσως ε, καλό θα ήταν να έχουμε αυτή τη φορά μια πιο ρεαλιστική στρατηγική για αυτούς τους στόχους. Αυτή είναι μια πρώτη ερώτηση. Μια δεύτερη ερώτηση τώρα. Και αφορά την κατάσταση στην Βόρεια Αφρική. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμμετέχει στις δράσεις μετά τις ε, συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική. Και η μετάβαση από τις ανθρωπιστικές δράσεις στην ε, προσπάθεια δημιουργίας χωρών, δημοκρατικών χωρών. Συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο και στη Λιβύη για το θέμα της ανάπτυξης τώρα και τη Συρία πέρα από την εξωτερική πολιτική και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που δεν συζητάμε ούτως ή άλλως εδώ στην Επιτροπή μας. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί το ρόλο της και τι ευθύνε της που είναι να προστατεύσει το λαό στη Συρία. Έχω διαβάσει ένα άρθρο ότι σταμάτησε να δίδεται η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ουσιαστικές σας ερωτήσεις, κύριε Μπέρμαν. Για την Κινέα Μπισάου με ρωτήσατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί φυσικά για την κατάσταση και έχει αναθεωρήσει τις κυρώσεις ούτως ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο ε, φάσμα φορέων. Εμπλέκεται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η κοινότητα των πορτογαλόφωνων χωρών που θα συζητήσουν αυτό το θέμα. Φυσικά γίνονται και συζητήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρξει δύναμη που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Το ίδιο φορά και την κατάσταση στο Μαλί, και, όπως και στην Κινέα Μπισάου. Εμείς ζητήσαμε, από το, ε, μας ζητήθηκε από το μηχανισμό ε, διευκόλυνσης της ειρήνης κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή η πρόταση δεν έχει λάβει, δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν για να δούμε πώ μπορούμε να ανταποκριθούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πάντω ένα θέμα βαθιά ανησυχία αυτό τη Γενέα Μπισάου. Και το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ. Υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθείτε θετικά, να δώσετε θετική απάντηση σε αυτό το αίτημα για ανάπτυξη δύναμη. Είναι θέμα συζήτηση του Συμβουλίου. Θα πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί καν η πρόταση. Δεν έχει διατυπωθεί καν η πρόταση πόσο μάλλον η απάντηση. Προσπαθώ να, σε, να σε εκμεύσω κάποιε απαντήσει. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ σε αυτή τη συνεδρία, όπω καταλαβαίνετε, λέει ο Δανό Υπουργό. Αλλά υπάρχει ανησυχία. Παρακολουθούμε το θέμα. Υπάρχει ένα γενικό αίτημα, α πούμε. Έχουν ξεκινήσει κάποιε συζητήσει, αλλά περιμένουμε ε, να διατυπωθεί πιο συγκεκριμένο αίτημα για να υπάρξει και απόφαση του Συμβουλίου για το, για το σημείο αυτό. Η έκθεση του ΩΣΑ δεν συζητήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου επίκειται ίσως σήμερα συναντήθηκα σήμερα το πρωί στην Κοπενχάγη ε, με τους αρμοδίους. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε να ε, ανταποκριθούμε στις ανησυχίες για το ODA για την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ξέρετε πώς ε, έχουν αυτά τα θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας και εταίροι. Είναι δύσκολο και για τον κόσμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήστε το και στις πρωτεύουσές σας παρακαλώ και στις χώρες σας. Ε, αυξήστε την πίεση και βεβαιωθείτε ότι θα στείλετε ένα μήνυμα για αυτά τα θέματα, και πόσο σημαντικά είναι και πόσο ζωτική σημασία για τον κόσμο ολόκληρο και για την Ευρώπη ειδικότερα. και η ύπατη εκπρόσωπο το θέτει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και συζητήθηκε και στο Συμβούλιο που το έθεσα εγώ. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη μεγάλη σημασία που έχουν αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη μεσού της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης θα πρέπει να διατηρήσει την ισχυρή της διεθνή παρουσία. Αυτό θα είναι και ένα μήνυμα για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Γιατί αν κοιτάξουμε γύρω μας, η ανάκαμψη της οικονομίας, η ανάπτυξη δεν έρχεται από την Ευρώπη, αλλά από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Και έχοντας μια διεθνή παρουσία η Ευρώπη, όχι μόνο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη μείωση της φτώχειας, αλλά θα αναπτυχθεί και η ίδια και θα δημιουργήσει θέση απασχόληση στην Ευρώπη. Και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το μήνυμα να το διαβιβάσουμε. Γιατί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μειώνεται σε ποσοστά. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε αυτό το μήνυμα πιο στεναρά και από κοινού. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι πολλές χώρες ε, στην Ευρώπη ε, δείχνουν ηγετική ε, θέση, αυξάνουν την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται και να εμπνεύσει και άλλες χώρες να προχωρήσουν. Κύριε Νόισερ, Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και πάλι. Για την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Okay. Εκτός μικροφώνου, κύριο κύριος Νόησερ δεν ακούμε τα σχόλιά του. Βεβαίως, θα τα διαβιβάσω αυτά στην κυβέρνησή μου και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ε, ε, η ατζέντα για την αλλαγή Βεβαίω, το τονίζετε μεγαλύτερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη. Και οπωσδήποτε θα μπορούσατε να πείτε ε, και να αντιτάξετε ότι η ε, υπόθεση του Συμβουλίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα μπορούσαν να είχαν ε, προχωρήσει περισσότερο. Υπάρχει όμως μια μεγάλη πλατφόρμα για την ατζέντα, για την αλλαγή, για να φτάσουμε σε μεγαλύτερα αποτελέσματα με μεγαλύτερο κοινό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Υπάρχει τώρα μια δέσμευση χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δωρητές να αναπτύξουν ε, μια ενιαία στρατηγική για την ανάπτυξη για να αυξηθεί η λογοδοσία, η προβλεψιμότητα σε μια χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ακόμα περισσότερα για να προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τις εταιρικές μας ε, χώρες. Αλλά και μεταξύ μας να συντονίσουμε το βηματισμό μας, να συγχρονιστούμε και με άλλες χώρες. Αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια λοιπόν όχι μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά όλες οι δωρήτριες χώρες με ένα κοινό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Αυτή είναι η ατζέντα για την αλλαγή και ε, υποστηρίζοντας ε, αυτά τα προγράμματα θα ε, υποστηρίξουμε και την κοινή συνεργασία στην Ευρώπη και το σχεδιασμό της. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες χώρες που συμμετέχουν πιλωτικά Θεοπία, Γκάνα, ε, Γουατεμάλα, Λάος και Ρουάντα ε, σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη γίνει και σε συνέχεια με το Νότιο Σουδάν ακολουθούν ε, Αφγανιστάν, Βερμανία και αργότερα το Μπαγκλαντές. Υπάρχει μια σειρά χωρών που αυτό μεταφράζεται σε πράξη, δοκιμάζεται, εξετάζεται και αναπτύσσεται περαιτέρω χρειαστεί. Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση που αναφέρατε. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνούν και τους τρόπους και τους δρόμους να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για κάποιες χώρες και να καλύπτουν όλο το φάσμα των σχέσεων μας με τις χώρες αυτές. Κοινά έγγραφα, πλαίσια και άλλη μια πλατφόρμα είναι αυτή Ξέρω ότι δείχνεται έτσι ανυπομονησία ως προς την ταχύτητα με την οποία προχωρούμε, αλλά γίνονται προσπάθειες για μια πιο κοινή προσέγγιση και κοινό σχεδιασμό, συνεργασία ε, και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. κυρία Κρέτσου. στον αναπτυξιακή στόχη της ε, χιλιετίας. Όπως σας είπα προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία, το είπατε και στην ερώτησή σας, θα πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στους στόχους της χιλιετίας. Δεν τους έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα και στο 2015. Δεν μπορούμε να τους ε, απεμπολίσουμε και να μπούμε σε μια νέα διαδικασία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προωθήσουμε με στένος και να εργοδοτήσουμε ε, για τους στόχους αυτούς ε, που έχουμε για τη χιλιετία μέχρι το 2015. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, ούτε χρονικά. Έχουμε μια τριετία ακόμα μπροστά μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την προσήλωση και το στένας μας αυτή. Αλλά βεβαίως να αρχίσουμε και συζητήσεις. Γιατί πολύ συχνά ε, αναφέρω πώς μπορούμε να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε τις φιλοδοξίες μας και να προσθέσουμε και άλλους στόχους, καινούριου στους στόχους χιλιετίας. Όπως σας είπα, η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε μια πρόταση για μια θέση της Ένωσης μετά το 2015. Στο αμέσως προσεχές μέλλον θα κατατεθεί αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ανάπτυξη σίγουρα θα συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και έντονα στο διάλογο. Όπω σα είπα προηγουμένω, διεθνώ έχουμε το πάνελ υψηλού επίπεδου. Τρει συμπρόεδροι, ο, Πρωθυπουργό Κάμερον του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρόεδρο Ούριο τη Ινδονησία και η Πρόεδρο τη Λιβερίας αυτοί οι τρεις έχουν ε, οριστεί. Οι υπόλοιποι μετά τη σύνοδο κορυφής ε, του Ρίου Συνήκωση και θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε το διάλογο για ε, τους στόχους μετά το 2015. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε και να αποσπάσουμε την προσοχή μας από τους στόχους της χιλιετίας μέχρι το 2015 που δεν έχουν όλοι υλοποιηθεί. Έρχομαι τώρα στην Αίγυπτο Βόρειο Αφρική. Όπως είπατε, βέβαια ορισμένα από αυτά τα θέματα υπερβαίνουν το πλαίσιο της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και πολιτικής, αλλά Στη Λιβύη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αποστολή που ολοκλήρωσε το έργο της για τη διαχείριση των συνόρων, για τον έλεγχο των συνόρων στη Λιβύη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Και εκτός αυτού, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω εγώ τι μπορώ να προσθέσω, ειλικρινά. Δεν έχω πλήρη εικόνα της προσέγγισης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Μπορώ να σας πω πολλά αν θέλετε για τη δανεική θέση για τη Συρία, για τα ανθρωπιστικά. Είμαστε σε στενή επαφή. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει κονδύλια και συμμετέχει πάρα πολύ στην ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και στην πρόσβαση στο εσωτερικό της Συρίας. Βέβαια, Σήμερα δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητική η κατάσταση σε σχέση με τις ανάγκες ή τις αρχές πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάντως, απομένει ακόμα πολύ δουλειά να γίνει και πιστεύουμε ότι παρότι έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά κάποιοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών στο εσωτερικό της Συρίας, αλλά θα πρέπει και οι ε, ε, τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό της Συρίας για τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Και αυτή η πίεση είναι πιο πιεστική παραποτέ και θα πρέπει να διατηρηθεί και να μείνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για αυτή τη συζήτηση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Του εύχομαι και καλό υπόλοιπο στην Προεδρία. Και μετά, βέβαια, καλές διακοπές που τις αξίζει κιόλα. Nous ε, Δεν μπορούμε να αρχίσουμε ακόμα τώρα την ψηφοφορία, γιατί τελειώσαμε νωρίτερα. Διακοπή λοιπόν τη συνεδρία μέχρι τι 5.30. Nous allons reprendre euh, après... Λοιπόν, α επαναλάβουμε μετά τη μικρή διακοπή για τις ψηφοφορίες. Αλλά επειδή σήμερα είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη ημέρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο πριν την ψηφοφορία στο Σαρλ Γκέρενς που έχει να μας πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι λίγο ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Θα ήθελα εισαγωγικά να σας πω την εξής μεταφορά. Η Επιτροπή μας είναι μια γέφυρα ουσιαστικά ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες εταίρους μας. Και η γέφυρα αυτή, όπως όλες οι γέφυρες, βασίζεται σε πυλώνες. Και από την άλλη εβδομάδα θα χάσουμε ένα πυλώνα που ονομάζεται Γκίδο Van να μην σας παρουσιάσω τώρα τη βιογραφία του, δεν είναι εύκολο. Είναι Βέλγος. Τι να κάνουμε, έχει καθένας το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Είναι Ευρωπαίος, ο καθένας έχει δικαίωμα να εξελίσσεται. Είναι μεταφραστής στο επάγγελμα, πράγμα που του επέτρεψε να καταλαβαίνει σε όλες τις αποχρώσεις τα διάφορα λόγια που ακούει δεξιά και αριστερά και μάλιστα πολλές φορές ψιθυριστά. Ε, και του οφείλουμε πάρα πολλά για τις διερευνητικές ε, αποστολές που είναι βάση της δουλειά μας. Έζησε πολλά χρόνια στην Αφρική. Ε, πράγμα που το καθιστά μάρτυρα της σημασίας των προβλημάτων που έχουν οι εταίροι μας. Το να το χαρακτηρίσει κανείς ευφυή είναι πάρα πολύ λίγο. Ο άνθρωπος είναι ε, ε, γάτος. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις ε, πόσο πολυμήχανος είναι, πόσο αποφασισμένος είναι, πόσο εργάζεται και πόσο ακούραστος είναι. Έχει και πολιτικές απόψεις, δεν τις έχει κρύψει ποτέ, αλλά αυτό ε, δεν τον απέτρεψε αυτό. είναι αμερόληπτος, ήταν στην υπηρεσία όλων των μελών της Επιτροπής, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύκτος. Γιατί βλέπουμε τι ώρα μας στέλνει τα email. Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Τι, να πει κανείς για τη ζωή του κύτου του οφείλουμε τόσο πολλά. Τώρα τι θα κάνει από εδώ και μπρο μετά την αποχώρηση του. Πρώτον αυτό δεν μας αφορά. Θα κάνει ό,τι θέλει. Ο Γκίδο αφού φύγει από εδώ είμαι βέβαιος ότι σίγουρα δεν θα ξεκουραστεί. Κάποτε είχε πει ο Φιντέλ Κάστρο ότι ένας καλός επαναστάτης δεν ξεκουράζεται ποτέ. Δεν πρόκειται να ξεκουραστεί λοιπόν. Άραγε είναι επαναστάτης ο Γκίτο. Όχι. Αλλά αυτό το γεγονό ότι δεν ξεκουράζεται ποτέ και το συνδέεται με το Φιντερελ Κάστρο είναι κάτι σαν επαναστάτης πάντως. Το 1968 ήταν μέσα στα πράγματα ακριβώς και κράτησε αυτό το πνεύμα να θέλει να αλλάξει τον κόσμο και ε, έχει βάλει και εκείνο το λιθαράκι του όπου ασχολήθηκε, βελτίωσε τα πράγματα. Δεν είναι επαναστάτης, αλλά είναι κάποιος ο οποίος βοηθάει να εξελίσσονται τα πράγματα. Και Έτσι λοιπόν στα γαλλικά όχι revolutionaire, evolutionaire, του λείπει το αρχικό ρο και δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Αυτά λοιπόν Γκίντο, εξ ονόματος εμού, βεβαίως προσωπικό, γιατί σε γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Είχε έρθει να με βρεις με τον ε, όταν ήσουν ε, διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του πριν από 10 χρόνια. Και πλέον κάποιος Βρετανός φίλος μου είπε μια μέρα δίνοντα τον ορισμό του φίλου το εξή. Φίλο είναι κάποιο τον οποίον σύναντά και μετά το χάνει για 10 χρόνια, 15 και μετά από 15 χρόνια Χωρί να εξηγήσει κανεί τίποτα στον άλλον, ξανασυναντιέσαι σαν να μην είχε χαθεί ποτέ. Και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει μετά από 10, 15, 20 χρόνια και να ζήσεις πολλά χρόνια και θα συνεχίσουμε να συζητούμε για τα ίδια θέματα. Σου οφείλουμε τόσα πολλά και δεν το λέω μόνο για μας, για μένα, εξ ονόματος μου προσωπικά, αλλά και εξ ονόματος όλων εδώ των ε, παρόντων και όλων εκείνων που είχαν ε, το προνόμιο να σε γνωρίσουν, να μοιραστούν λίγο από το δρόμο σου μαζί σου και μπορεί να είναι περήφανοι που σε συγκαταλέγω μεταξύ των φίλων τους, γιατί είσαι πραγματικά πολύ σπουδαίος. Ε, Γκίντο, ευχαριστώ και πάλι. Καλή τύχη. Θα είμαστε πάντα εδώ για σένα και είμαι βέβαιος ότι θα ε, ακούσουμε ε, ξανά ε, να μιλούν για σένα γιατί σίγουρα δεν ξεκουράζει. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ συγκινητικά αυτά του Σαλ, δεν πρόκειται εγώ να πω τίποτα, τα κάλυψε όλα. Αλλά ως εισηγητής ε, για το σημαντικό μέσο DCI το, ε, ε, πρέπει να σου πω ότι θα μου λείψει πολύ. Εγώ θα το 7 στην Επιτροπή αυτή ή το 8 δεν θυμάμαι και μου έκανες μια εισαγωγή πάρα πολύ σημαντική για μένα και σε ευχαριστώ. Είσαι από εκείνους που πιστεύουν στην ανάγκη και την ανάγκη, όχι τη δυνατότητα, στην ανάγκη ενός κόσμου που να βασίζεται σε αρχές, σε αξίες και περισσότερο από τα πεζά της αγοράς ή του χρήματος και ίσως στην Επιτροπή μας αυτό είναι πολύ πιο ε, αναγκαίο από ό,τι άλλες επιτροπές και είσαι στη σωστή θέση. Κρίμα πάρα πολύ που φεύγεις θα τι να κάνω, θα προσπαθήσω την έκθεση μου να την ολοκληρώσω. Θα μας λείψεις ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις που είναι πολλές φορές επίπονες με το Συμβούλιο γιατί οι σχετισμοί δυνάμεων ε, Συμβουλίου Κοινοβουλίου ήταν κάτι που γνώριζες με τέτοιες λεπτομέρειες και με τόσο καθαρό τρόπο ήξερες και την τελευταία απόχρωση. Θα προσπαθήσω ε, να συνεχίσω με το διάδοχό σου που είναι πάρα πολύ άξιος, πάντα ήσουν στο πλευρό μας. Σκεφτόμασταν πάντα ότι είσαι πιο έξυπνος από μας. Ε, για, καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο, αλλά πάντα όταν είσαι συνεργάτης ενός ευρωβουλευτή πρέπει να του δίνεις ε, την εντύπωση και να ε, μην τον αφήσει ποτέ να καταλάβει ότι είσαι εσύ πιο έξυπνος από εκείνον. Ε, παρακαλώ να παραμείνεις και στη διάθεσή μας και με βέβαιος και με τη Μαρίκα και με τα email που θα επικοινωνούμε για να μας βοηθήσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much, President. I'd like... Ευχαριστώ. Όπως και οι προλαλήσαντες και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή σύνταξη στον Κίντο. Είναι μια πολύ ειδική περίσταση αυτή. Μέσα με τα χρόνια έμαθα πόσο επιδέξιος είναι ο Γκίντο και στην πολιτική χρειάζεσαι τέτοιους βοηθούς, χρειάζεσαι ανθρώπους που ξέρουν πώς λειτουργούν τα πράγματα και που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρόνο και ενέργεια για πολλά πράγματα. Έχουμε εισηγητή στο πρώτο DCI. Ε, ήταν η πρώτη μου θητεία στο Κοινοβούλιο. Ήμουν υπουργό εξωτερικών υποθέσεων αλλά τότε συγχωνεύαμε 16 κανονισμούς σε ένα. Ποτέ στην πολιτική μου καριέρα δεν είχα αισθανθεί αυτή την πίεση που αισθάνθηκα εκείνα τα δυόμιση χρόνια για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό στο Κοινοβούλιο. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια ο γραμματέας αυτής της Επιτροπής υπό την αιγύδα του Γκίντο με καθοδήγησε πολύ επιδέξια. Ήταν μια μεγάλη παρατηταμένη περίοδο, δυόμιση χρόνια όπως σας είπα, και εκείνο ε, ήταν ε, συνέχεια παρόν. Με κατέπληξε πραγματικά. Δεν θα είχα μπορέσει να συμμετάσχω σε όλες αυτές τις συζητήσεις ε, χωρίς τη συμβουλή του. Πάνω απ' όλα όμως θα μας λείψει γιατί πάντα εξέφραζε το κοινοβούλιο και το υπερασπιζόταν. Δεν συνειδητοποιούμε πάντα πόσο επιδέξια είναι τα άλλα δύο θεσμικά όργανα εμείς έχουμε μια τάση να εμφανιζόμαστε διαιρεμένοι και να παρουσιάζουμε το πάθεια. Και νομίζω ότι η μεγάλη δύναμη του Γκίντο είναι ότι εξέφρασε τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Ήμουν εισηγητής και πάντα να ζητούσα την συμβουλή του όπως και άλλοι εισηγητές, άλλοι συντονιστές κτλ. Και σου είμαστε ευγνώμονες, ε, Καλή τύχη σε ό,τι κάνει. Ε, να είσαι πάντα σε επαφή μαζί μα, όχι ε, στι 3 και 4 ώρα το πρωί βέβαια, αλλά πάντα θέλουμε να κρατήσουμε, να έχουμε μια επαφή μαζί σου. Ο κύριο Ντέβα ζητάει τον λόγο. Ε, you, like to... Ευχαριστώ. Μέχρι πριν 10 λεπτά η μέρα μου πήγαινε καλά. Ήμουν άνετος. Και τώρα όμως άκουσα αυτή την κατακλυσμιαία ανακοίνωση ότι ο Γκίντο εμφανίζεται εδώ μαζί, είναι εδώ μαζί μας για τελευταία φορά, είναι τελευταία του συνεδρίαση. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά θέλω να πω ότι ο Γκίντο είναι πάνω απ' όλα κύριος. Και είναι πολύ δύσκολο τη σήμερα ημέρα να βρει κανείς ένα πραγματικό κύριο. Ήταν ευγενής, μας βοηθούσε και όταν λέει όχι σε κάτι, τον ευχαριστείς γι' αυτό. Αυτή είναι η ουσία του Κυρίου. Ελπίζω να περάσει καλά τη σύνταξή του. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Φαντάζομαι θα ασχοληθεί με την Κυπουρική. Ναι, γνέφει ο Γκίντο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σου, για τις συμβουλές σου, για την ευγένειά σου και τις γνώσεις σου. Με καθοδήγησες με τέτοια επιδεξιότητα σε αυτόν τον ε, λαβύρινθο το θεσμικό, όπου οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά παρόλα αυτά οι αξίες παραμένουν. Εσύ ήσουν πραγματικός πυλώνας, απαρασάλευτος. Ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής, να ευχαριστήσω τον Κίντο για την τεράστια προσπάθεια που έκανε για την Επιτροπή μας και για την ε, υποδοχή που μου επεφύλαξε όταν έφτασα εδώ το 2009. Έκανε ό,τι μπορούσε, ούτω ώστε αυτή η Επιτροπή να συνεχίζει να εργάζεται παρά την ε, ασχετοσύνη της Προέδρου της. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι καλή σύνταξη όπου πας. Είμαι σίγουρη θα συνεχίσει την προσπάθεια ούτω ώστε οι σχέσεις βορρά-νότου να είναι πιο ισορροπημένες και να μειωθεί η φτώχεια. Γεια σου και μην μας ξεχνάς. Εδώ κανονικά ένας γραμματέας δεν μιλάει σε συνεδρία επιτροπής γιατί είμαι διοικητικό υπάλληλο και τώρα παραβαίνω όλους τους κανόνες. Προσπάθησα πάντα να είμαι σωστό υπάλληλο και να τηρώ τους κανόνες. Αλλά πώς να σας εκφράσω πόσο συγκινημένος είμαι. Θέλω να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, με τα εγγόνια μου στην Νικαράγουα, Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να φύγω από εδώ, από αυτή την Επιτροπή. Να φύγω από σας. με τους οποίους αντίθετα από ό,τι συμβαίνει αλλού ε, είχα μία σχέση έτσι στενή. Ήμασταν μια ομάδα, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει αλλού. Είμαστε μια ομάδα με την ίδια αποφασιστικότητα και τους ίδιους στόχους. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την αποφασιστικότητά μας, με αποφασιστικότητα αυτόν τον αγώνα. Δεν θα είναι εύκολο. Εγώ τώρα θα είμαι στο περιθώριο και θα παρακολουθώ απλώς τα τεκτενόμενα μέσα από το web streaming, ό,τι συμβαίνει σε αυτή την επιτροπή. Ε, συχνά μπορεί να λέω, α, Θεέ μου, γιατί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, λάθος κάνουν. Το τελευταίο χρόνο σας έχω δώσει και το δικό μου προσωπικό email και ελπίζω από καιρούς καιρό να παίρνω νέα σας. Και όποτε είμαι στο Βέλγιο με τη γυναίκα μου, θα είμαι πίσω στην, στα καθίσματα των Κροατών για να βλέπω πώς υπερασπίζεται τις αξίες μας αυτή η Επιτροπή ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για όλα και καλή τύχη και σε όλους σας. Ε, θα, κάνουμε, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, αλλά πρώτα θα κάνουμε ε, μία δοκιμή. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Θα υπερψηφίσουμε. Βλέπω τρεις-τέσσερις δεν έχω έχουν ψηφίσει. Ε, 21 ψήφισαν ενώ συνήθως είμαστε 24. Δεν έχω μαζί την κάρτα μου. Με συγχωρείτε. Θα σας σημειώνουμε λοιπόν. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν δύο ακόμη οι οποίοι δεν έχουν ε, ψηφίσει. Έχουν ξεχάσει τις κάρτες τους. Δύο ακόμη άτομα δεν έχουν ψηφίσει. Τώρα όμως είμαστε εντάξει. Λίγοι. Ψηφίζουμε λοιπόν την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Γκάι Μίτσελ, πρώτη τροπολογία. Τροπολογία 1 έως 6. 1 έως 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 έως 10. Ψηφίζουμε από κοινού το 7 έως 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ε, ομόφωνα 25 υπερψήφισαν. Τώρα θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση της κυρίας Ζήμερ. Ε, έχουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και ψηφίζουμε και την ε, γρομοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. Οι 13 υπέρ, 8 κατά και 4 αποχές και εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Γκερέρο Σαλόμ και έχω να σας ανακοινώσω δύο πράγματα. Στην προφορική τροπολογία 4, στο εκτιμώντας 14, η τροπολογία της κυρίας Νίμπερα Στραμ ε, αγγλικά πρέπει να λέγει coherence και όχι cohesion. Και μετά, όσον αφορά την τροπολογία 5 του εισηγητή, η τροπολογία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν έχει περιληφθεί εκ παραδρομής στον κατάλογο ψηφοφορίες και προτείνω να το ψηφίσουμε πριν από την τροπολογία 6 του εισηγητή. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 18. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη. 17 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 που δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 23 λίγη εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά λίγη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 αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. Προφορική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την γνωμοδότηση όπως άλλαξε και ε, ξεκινά η ψηφοφορία ε, λίγη 22 υπέρ, άρα κρίθη. Ψηφίζουμε τώρα τη γνωμοδότηση του κυρίου Κασμάρεκ. Τροπολογία 1 υπέρ. Πρόεδρε, ε, μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ μέχρι την 26 λέει ο κύριος Μίτσελ. Μέχρι 25, συγγνώμη. Όλες μαζί από την 1 μέχρι και την 25. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε, αμού. Όχι. Καλά. Ο κύριος Ντόνσκης. Μέχρι την 22, ναι, 25 δεν θα μπορέσω, λέει ο συντάκτης των τροπολογιών μέχρι και την 22, εντάξει. Ωραία. 1 έως και 22 με τη σειρά αυτή, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 επίσης 26 ε, ψηφοφορία κατά τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Άποχες. Εγκρίνεται. Κύριε Μίτσελ, μπορούμε να ψηφίσουμε και πάλι ομού κάποιες τροπολογίες. Ποιες θέλετε όμως. Μέχρι πού. 28. Όχι, δεν γίνεται. Μέχρι πού. Πώς θέλετε να το χωρίσετε κύριε Μίτσελ, ποιες τροπολογίες να ψηφίσουμε μαζί. Μέχρι τη 10. Μέχρι τη 10. Συμφωνείτε. 8, 9, δηλαδή 27, την προφορική και τη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία παριθμών 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε τώρα τη γνωμοδότηση της Φιώνα Χολ. Η τροπολογία 29 ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία έρθουν 4 είπε. Τριάντα δύο. 32 κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία βαρθών 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία βαρθών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. το τροπολογία υπερθών 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 38 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται η τοπολογία μόνο 8 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται ή 39. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Καλώς. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 39. Le vote σε adopted. Ναι. adopted. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Ερχόμαστε στη 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ouais, je vérifie. Je n'ai pas vu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 αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ Η 45 εγκρίθηκε, οπότε η 17 καταπίπτει και τώρα ψηφίζουμε τη 18. Υπέρ. 18. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα. Έχουμε την προφορική παρθόνα 1 υπέρ. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας 1. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Qui Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία στη συνέχεια επί του συμβιβασμού 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχο θέλετε καλώς άρχιτε ψηφοφορία Le vote est clos. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Euh, compromis 1, Η συμβαστική 1 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Ψήφοφορία κατά τμήματα.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 Λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Στην 27. 27. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Τσεκ. Ωραία, ελέγχουμε την 27. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να το ελέγξουμε. Le Πέρας. Α, εγκρίθηκε, συγγνώμη, έκανα λάθος. Η τροπολογία παριθμό 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο. Α, κύριε Χόλ. Με ένα-δύο άτομα θεωρούν ότι δεν ψηφίσαμε τροπολογία 5. Η γραμματεία μπορεί να τσεκάρει αν ψηφίσαμε ή όχι. L'amendement Thank you. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Είναι η τελική ψηφοφορία. Το κειμένο που τροποποιήθηκε. Πέρας ψηφοφορίας. Υπερψηφίστηκε. Πέρασε με 24 ψήφους. Και τώρα πάμε στη δεύτερη γνωμοδότηση της κυρίας Φιώνα Χολ. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Ε, πρώτη προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την πρώτη προφορική τροπολογία. ψηφίζεις εσύ. Δεν βλέπω το... με το καρτελάκι σου και τι ψηφίζεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία ακόμα. Γιατί... Λοιπόν, Υπάρχουν δύο άτομα που δεν ψήφισαν. Ακόμα ένας. Bon, euh, voilà, vote Ωραία, πέρας ψηφοφορία. Υιοθετείτε. Euh, Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 3 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Υπέρ, ξανά, της πρώτης τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. Πέμπτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε... Euh, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα, ψηφοφορία, Υιοθετείτε. Oui adopté. Et donc, nous allons maintenant voter l'opinion. Ψηφίσουμε τώρα τη γνωμοδότηση. Ηλεκτρονικά. Όπως έχει τροποποιηθεί. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται. Alors, Ψηφίσουμε την έκθεση του Γιάν Σαραντίλα. Έχετε το λόγο. Ένα διαδικαστικό σημείο θέλω να θέσω εδώ. Η κυρία Ζαρα... δεν είναι εδώ. Θέλουμε να μην ψηφίσουμε τον κύριο, την ε, έκθεση του κυρίου, η οποία απόφαση θα αναθεωρηθεί με βάση τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμβατότητα της ε, συμφωνίας κατά των απομιμήσεων με τη συνθήκη. Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι σαν γι' αυτό το κείμενο όταν ξέρουμε ότι εκρεμεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το αν η νομοθεσία μας συνάδει με τη συνθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία μέχρι να δούμε τι απόφαση θα πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να δούμε αν είμαστε συμβατοί. Το κείμενό μας δηλαδή είναι συμβατό με τις συνθήκες. Μπέρμαν. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την πολιτική μας άποψη για την άκτα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία. Και σε άλλες ε, επιτροπές έχουν ήδη ψηφίσει εξάλλου. Madame Stifler. Non, non, mais j'allais dans le même. Αν ψηφίσει η ΙΝΤΑ, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, τι νόημα έχει να, πούμε, να αποφασίσουμε εκ των υστέρων. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αυτό το διαδικαστικό σημείο καταρχήν. Ποιο είναι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας. Ποιο είναι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται το διαδικαστικό έτοιμο του κύριου Ντέβα για καθυστέρηση πληροφορίας, αλλά θα ψηφίσουμε. Πρώτο συμβασμός. Ένα έως τρία. Ψηφίζουμε μαζί. On block. Υπέρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qui est contre. Κατά. Qui, qui s'abstient. Αποχές. Donc, les, les compromis... Οι συμβιβασμοί 1 έως 3 υιοθετούνται λοιπόν. On block. Και τώρα επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ouais. Πέρα ça c'est Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Με επαρκή πλειοψηφία. Μεγάλη πλειοψηφία. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία που γίνεται ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε. Encore. Euh, Presidenta, Presidenta. Oui. D'accord. Alors, Alors, comme il manque toujours une voix qui a une demande de clarification, on va recommencer le contrôle. Μου λείπει μία Ε, θα ξαναρχίσουμε τον έλεγχο αφού πάρετε το λόγο. Ouais. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Πρόεδρε, είχαμε πρόβλημα εμείς με το κατάλογο ψηφοφορία μας και θα παρακαλούσα να ε, επαναλάβουμε αν γίνεται τις δύο τελευταίες ψηφοφορίες. Έχουμε ένα πρόβλημα ε, εκτύπωσης του κατάλογου ψηφοφορία μας. Να επαναλάβουμε τις δύο ψηφοφορίες παρακαλώ. Berman, vous avez demandé la parole. Vous voulez la parole, Monsieur Ναι, υπάρχει λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας μας. Ε, εμείς θέμε. Θα ξαναψηφίσουμε. Όλες τις τροπολογίες. Γιατί είναι ίδιες. Όλες τις τροπολογίες μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Το κάνουμε ηλεκτρονικά. Για να μην κάνουμε λάθος. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 1 έως 3 και τους τρεις μαζί. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Voilà. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση, όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε τώρα.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

της Επιτροπής μας για το MIFID και το MIFIR. Δηλαδή, το πρόγραμμα της ΕΚΟΝ, ε, το πιο σημαντικό αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Πρόκειται για δύο κείμενα που θέλουν να περιορίσουν, να εξαλείψουν την κερδοσκοπία στις πρώτες σύλλες. και προτείνω 60 τροπολογίε. Ο στόχο μας είναι να δώσουμε ορισμό της κερδοσκοπία, της υπερβολικής και αχαλίων της κερδοσκοπία. και να ενισχύσουμε την εξουσία των ελεκτικών μας αρχών και φορέων στις αγορές. Γιατί ξέρουμε ότι η κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες οδηγεί σε μία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών εντελώς ανώφελα και περιτά. Και έχει σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες γιατί επηρεάζει και τις τιμές των τροφίμων. Το κόστος ζωής βεβαίως επηρεάζει και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε και να περιορίσουμε την κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες. Σε σχέση λοιπόν με το κείμενο της ε, Κομισιόν, έχω να πω ότι δεν υπάρχει ορισμός αυτής της υπερβολικής κερδοσκοπίας. Εγώ στην ε, τροπολογία 14 της MIFID προτείνω έναν ορισμό της υπερβολικής κερδοσκοπίας. Θέλω οι εξαιρέσεις των κανόνων να περιοριστούν οι εξαιρέσει από τους κανόνες και οι έλεγχοι να αφορούν όλους τους φορείς που παρεμβαίνουν στην αγορά. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω τον νόμο Dodd Frank τις ε, εξαιρέσεις που, ε, στις οποίες επανήλθαμε από την κρίση του 2008. Στο κείμενο της Κομισιόν δεν υπάρχει η μέγιστη θέση. Επίσης δεν προσδιορίζει τι είναι αγώνας κατά της κερδοσκοπίας και δεν λέει ότι είναι ο στόχος μας ε, με σκοπό την καλή λειτουργία της αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα όρια θέσεων στο άρθρο 59 του κειμένου της Κομισιόν και στην τροπολογία μου 14 ε, και στις επόμενες θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Εν συνεχεία, στο κείμενο για το MIFIR, για τον καονισμό δηλαδή, για τις αγορές, θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα, ε, ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών στα άρθρα 31, 32 και 35. Και εκεί έχουμε τις ε, σχετικές τροπολογίες 1 με 20. Πρόκειται λοιπόν για δύο κείμενα που έχουν τεράστια σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο και την αιτιολογική σκέψη και να δείτε και τις 60 τροπολογίες. Έχετε προθεσμία για την κατάθεση και άλλων τροπολογιών μέχρι αύριο. Τι ώρα όμως, μεσημέρι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι νομίζω. Ακριβώς, αύριο μέχρι τις 12, λοιπόν. Ο κύριος Μίτσολ ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για, αυτό το, για αυτή την πολύ σημαντική γνωμοδότηση. Είναι μια πολύ σημαντική για τις ε, χρηματοοικονομικές ε, υπηρεσίες διότι πρέπει μετά την κρίση να προσαρμοστούμε και να προβούμε σε μια μεταρρύθμιση κατόπιν των πολλαπλών νομοθετικών προτάσεων που εξετάζονται στην Επιτροπή Οικονομικών που δραστηριοποιείται στον τομό αυτό πρέπει η ΔΕΒΕ να αποφανθεί για την ΜΥΦΙΤ ε, και ιδίω ε, διότι και το θέμα των πρώτων υλών στις υποανάπτυξη χώρες είναι πολύ σημαντικό και πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Όσον αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές που επηρεάζουν την αστασή, δεν μπορούμε να ε, ελέγξουμε τις κλιματικές συνθήκες αλλά η πληροφόρηση στην αγορά ε, και ε, άλλες δυνατότητες είναι μέσα στο πλαίσιο του εφικτού και έτσι θα μπορούσαν οι ρυθμιστές να ρυθμίσουν την κρίση και ιδίως τις εχμές της προς τα πάνω ή προς τα κάτω και ε, θα ήθελα σαν σαν σκιώδης εισηγητής και συντονιστής του ΕΛΚ να πω το παρακολουθώ εκ του σύνεγγης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Τερέζα Φαμπρέγκα Φερνάντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Υπουργός. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σκοπεύει να ε, ασχοληθεί με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα για να βελτιώσει τη διαφάνεια, να μειώσει τις εξαιρέσεις και να δούμε πώς μπορεί το θέμα αυτό να παρακολουθηθεί καθώς συγχρόνως και να προταθούν εναλλακτικές λύσεις βλέπουμε ότι αυτό αναφέρεται στις συστάσεις του G20 και ακολουθώντας τις βλέπουμε ε, ποιες είναι οι δυνατότητες ε, ιδίως συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες όπως ανέφερε η συγγήτρια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρχει σαφήνεια σε αυτές τις τροπολογίες για να μην μπορεί κανείς να παρατα... Ε, παρακάμψει αυτές τις προτάσεις και χαιρετίζουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ότι θα ε, επανέλθετε στους περιορισμούς της Αμερικής και ελπίζω ότι θα πορευτούμε όλοι μαζί. Οπότε, η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 18 Ιουνίου από τις 15 ε, έως 18 και 30 και 19 Ιουνίου από 9 έως 12.30 και 15 με 18.30 σας ευχαριστώ και λύεται η συνεδρίαση.